Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζονται οι εργασίες μα. Ε, η μερίσια διάταξη. Δεν έχω ε, ακούσει να θέλετε αλλαγέ, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Στο 2 σα παραπέμπω στα cont news και τι γλώσσε που έχουμε σήμερα στη συνεδρίαση. Κατά τα άλλα, δεν έχω να σα πω τίποτα. Ε, Όπω πάντα, παγκοσμίω μπορεί να μα παρακολουθεί ο κόσμο ε, στο διαδίκτυο. Παρακαλώ, ετοιμάστε ε, τις κάρτες ε, ψηφοφορίες σας, γιατί έχουμε τώρα το σημείο 3 που είναι ψηφοφορίες και θα τις χρειαστούμε πολέμηση της απάτης. Ο κύριος Σαλαφράνκα είναι ο συνάδελφος εισηγητής. Έλετε το λόγο κύριε Σαλαφράνκα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Ε, Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά με τους συναδέλφους των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ε, θέλω να σας πω μόνο ότι στις πρώτες τροπολογίες 44, 45 και 36 δεν μπόρεσα να τις υποστηρίξω. Όχι επειδή διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά γιατί είναι εκτός τόπου τώρα. Δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο. Αλλιώς ε, με τα χαράς δεν έχω κανένα πρόβλημα, καμία δυσκολία, αλλά δεν είναι ε, του παρόντος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για να ψηφίσουμε, πιστεύω. Ε, ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. 44. Υπέρ. Κατά. Ξανά, λοιπόν. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αχα αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές. Τώρα μόνο υποθέσεις και κασίες μπορώ να κάνω για το πώς ψηφίζουν οι διάφορες ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές. Ας το κάνουμε ηλεκτρονικά για να ξεβερδέψουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 7. Τώρα το βρήκαμε. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά θα το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Την 11 παρακαλώ. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά για καλό και για κακό. Δεν καταλαβαίνω τους συσχετισμούς σήμερα το πρωί. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 ε, του προπολογισμού δεν ψηφίζεται. Πάμε στην τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 επέ κατά αποχές. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό ηλεκτρονικά, 14. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά Μπορούμε να την ελέγξουμε σας παρακαλώ την 27. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 31 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, το 31. Πέρας. Απορρίπτεται 32 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά απόχε εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 35 κατά πίπτη. Η ένα του προπολογισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 του προπολογισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτς 3 δεν την ψηφίζουμε, 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά αποχές Μπορούμε να την ελέγξουμε αυτή ηλεκτρονικά, σας παρακαλώ, την 37. Πέρας εγκρίνεται. Ε, μπάτς 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε αρχίζει ψηφοφορία ε, ονομαστικά και ηλεκτρονικά. Γνωμοδότηση καλύτερα. 17-0 εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά μου. Και ερχόμαστε στην επόμενη γνωμοδότηση για την κοινή πολιτική και τον αντίστοιχο κανονισμό. Ε, η κυρία Σμίτ είναι συντάκτρες νομοδότησης, επιθυμεί το λόγο όχι, οπότε και θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές. Ε, μήπως μπορούμε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Το δεύτερο τμήμα τη τροπολογία παρελθόν 16, έλεγχο παρακαλώ, επαλήθευση. Ε, ολοκληρώθηκε επαλήθευση, ο έλεγχο και απορρίπτεται. Η 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 19 υπέρ, κατά, αποχές. Μήπως μπορούμε να ελέγξουμε 19. Απορρίπτεται το 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ε, μπορούμε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Το 20 το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27. Σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, ε, αποχές. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ, επαλήθευση. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η υπεριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 31 με προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 33 με προφορική τροπολογία, ε, καμία αντίρρηση, καμία διαφωνία, υπέρ κατά ε, επαλήθευση παρακαλώ για την 33. έλεξε η επαλήθευση. Δεκτή. Yeah. Ε, μισό λεπτό. Υπαριθμόν 2. Υπέρ. Η 3 αποσύρθηκε. Η 4. Υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε για την 4 παρακαλώ. Και η 2 είχε αποσυρθεί. Η 4 επαληθεύουμε για τη 4. Δεκτή η 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 35 καταπίπτει. Η 7 αποσύρεται. Η 8 επίσης. Η 36 υπέρ κατά μπορούμε να ελέγξουμε την 36. Έληξε η επαλήθευση. Η 9 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 13 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να έχουμε επαλήθευση για την 13 παρακαλώ. Νομίζω ότι έγινε δεκτή, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Απορρίπτεται με ισοψηφία η 37 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, η 14 ε, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Η 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή ονομαστική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Συγχαρητήρια για αυτή τη δύσκολη δουλειά. Πάμε τώρα στην γνωμοδότησή μας για το στρατηγικό σχέδιο, ε, το Ταμείο Εγγυήσεων και την Ήπετρο, εισηγητής ο κύριος Τσέλερ, ο οποίο δεν είναι εδώ, ω εκ τούτου δεν μπορεί να λάβει και τον λόγο, δεν έχει ορίσει και αναπληρωτή. Α ψηφίσουμε λοιπόν. Η 11 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχέ, δεκτή. Η 12 υπέρ, κατά, αποχέ, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 12. Και έγινε δεκτή. Η 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 14, υπέρ, κατά, αποχές, μήπως μπορούμε να ελέγξουμε την 14. Δεκτή. Η 15 υπέρ, κατά αποχές δεκτή η 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 20 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά καλύτερα να ελέγξουμε παρακαλώ για την 20. δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 24 παρακαλώ γιατί νομίζω ότι έχει γίνει δεκτή αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Για την 24 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πράγματι δεκτή, 24 δεκτή, 25 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 26 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 27 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 28 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 31 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεκτή, 33 υπέρ κατά για την 33. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Απορρίπτεται. Was sagt die Geschäftsordnung zum Wrong Button? Ja, normalerweise ändert der Πρόεδρος, ε, κατά κανόνα το wrong button δεν αλλάζει την ε, ψηφοφορία ε, και δεν θέλω τώρα να σχοληθώ με τον κανισμό, γιατί και εσείς είσαι τόσο συμπαθητικός Αυτός είναι και ο κίνδυνος που υπάρχει στο επάγγελμά μας δεν μπορώ να κάνω καμία εξαίρεση. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι που ήμασταν. 33 απορρίπτεται η 34 υπέρ, κατά, αποχές και εδώ ε, για την 34 παρακαλώ. Απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές ε, δεκτή, 37 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 36 υπέρ κατά αποχές, ε, μήπως να κάνουμε επαλήθευση για την 36 παρακαλώ. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. Οι 38 και 39 είναι ταυτόσημες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Και εδώ παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση για την 38 και την 39. Δεκτή και οι δύο δεκτές. 40-41 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 42-43 υπέρ, κατά αποχές δεκτές, 44-45 υπέρ κατά αποχές δεκτές, οι 2 και οι 46 υπέρ κατά αποχές δεκτές, οι 47 και οι 48 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτές, οι 49 υπέρ κατά αποχές, ε, μήπως μπορούμε να ελέγξουμε γιατί οι 49 Ολοκληρώθηκε η επαλήθευση. Απορρίπτεται η 50 υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση και για την 50. Λυπάμαι. Απορρίπτεται. Η 51 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται η 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 58 σε δύο τμήματα, ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, Μπορούμε να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Απορρίπτεται. Η 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 60 με προφορική τροπολογία δεν έχει κανείς αντίρρηση. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 63 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 63. υπέρ κατά 65, ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η, 70 ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Δεκτή. Η 71 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η 72 υπέρ κατά αποχές ε, ε, να ε, κάνουμε επαλήθευση για την 72 παρακαλώ. Δεκτή. Πάμε στην 73. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτή. 74. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 74. δεκτή. Η 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 80 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η 81 υπέρ κατά αποχές ε, Η 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 84 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 86 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 87 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές. Ε, μήπως μπορούμε να ελέγξουμε την 6. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. απορρίπτεται. Η 91 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, η 92 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, η 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 7 υπέρ κατά ε, πρέπει να ελέγξουμε την 7. Την 7 παρακαλώ. Λοιπόν, υπέρ. Η 8 υπέρ <laughs> κατά αποχές ε, δεκτή. Η 96 καταπίπτει, η 97 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές δεκτή, η 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και η 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έτσι λοιπόν η γνωμοδότηση έγινε δεκτή, εγκρίθηκε με αποτέλεσμα 19 υπέρ 1 κατά. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Πάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 5 στην ημέρηση. Ωραία, τα βρήκαμε και μπορούμε να προχωρήσουμε. Το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη, οι έρευνε ε, του Γραφείου για την Καταπολέμηση της Απάτης, Όλαφ, ώψη και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ε, η αποδοτικότητα του και αποτελεσματικότητα είναι συναπόφαση αυτό το θέμα, η συγγήτρια υποφαινόμενη. Έχετε την έκθεση περίπου 108 με 110 τροπολογίες υπάρχουν. Θα συζητήσουμε κάτι λιγότερο από μία ώρα. Θέλω να καλωσορίσω το Γενικό Διευθυντή ε, της όλα τον κύριο Ήταλα, και το επίτελείο του. Καλωσορίσατε. Ε, και ε, όπως μπορείτε να δείτε από την έκθεση, ασχολήθηκα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό της Όλαφ και συμφωνώ σε γενικές γραμμές. Θυμάμαι πολύ καλά την περασμένη αναθεώρηση που ε, διήρκησε μία έπτα αιτία. Ελπίζω αυτή τη φορά το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να τα καταφέρουν κάπως νωρίτερα, γιατί ε, έχει ήδη προγραμματιστεί αρκετά γρήγορα μετά τις ευρωεκλογέ να αρχίσουμε τριμερείς διαπραγματεύσεις, τον τριμερή διάλογο. Το σχέδιο εκθεσή μου υποστηρίζει ε, την ε, πρόταση προσαρμογής στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καλωσορίζω και τα διδάγματα που βγάλαμε από την αξιολόγηση το 2017. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αξιολόγηση ε, για τις δικές μου προτάσεις, γιατί ακριβώς οι περισσότερες από αυτές βασίζονται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Πού κατέληξε η αξιολόγηση ότι η αποτελεσματικότητα των ερευνών Τη ε, της ΟΛΑΦ πρέπει να αυξηθεί. Πώς θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν για τους επιτόπιους ελέγχους στα κράτη-μέλη, ε, αλλά και να απλουστεύεται η πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Το είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το καλωσορίζω και εγώ. Επίσης, καλωσορίζω διευκρινήσεις και απλουστεύσεις ε, ό,τι φορά τη διαδικασία. Το έχουμε συζητήσει σε διάφορα εργαστήρια, βέβαια τίθεται το ερώτημα αν αρκεί η πρόταση αυτή για να είναι εγγυημένη η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ιδιαίτερα να έχουν κάποια χρησιμότητα τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της Όλαφ όταν ε, θα αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλυσε τα προβλήματα. Και επίσης πιστεύω ότι για τα διδάγματα που έχουμε ε, ξέρω για το παρελθόν χρειάζεται κάποια βελτίωση, χωλαίνει ακόμα υπόθεση. Συνοψίζω. Έχω κάνει κάποιες διευκρινήσεις και λεπτές ρυθμίσεις σε σχέση με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχω ζητήσει απλούσευση των διαδικασιών και καλύτερη συνέχεια να δίνεται στα αποτελέσματα από τα κράτη-μέλη. Ε, γιατί αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα ε, με τις δικαστικές διαδικασίες, γιατί κάνει η όλαφ και τα δικαστήρια στη συνέχεια ε, δεν δίνουν συνέχεια. Θυμάστε μια φασαρία που έγινε, δεν την έχω ξεχάσει ούτε κι εσείς, για την πρόσβαση στα έγγραφα, ποιος παίρνει ποια έγγραφα και ποιος δικαιούται τι. Και πάντα τα δικονομικά δικαιώματα των εμπλεκομένων προσώπων είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίσης καταργώ τη διάκριση εσωτερικής-εξωτερικής έρευνα. Καλά δεν είναι ίσως η πιο χτυπητή αλλαγή, ε, αλλά για λόγους τεχνικούς έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες, ιδιαίτερα τα άρθρα 3 και 4. Οι επιπτώσεις όμως είναι μάλλον περιορισμένες. Έχω διαγράψει κάποιες ε, διπλές επικαλυπτόμενες νομικές ρυθμίσεις και κείμενα. Υπάρχουν πολλοί ε, λόγοι και καλοί λόγοι για την κατάργηση τη διάκριση αυτή σε εσωτερικέ και εξωτερικέ έρευνε. Το είπαμε και την περασμένη φορά σε διάφορα εργαστήρια. Δεν έχουμε προχωρήσει στι διαπραγματεύσει. Γιατί να καταργηθεί αυτό. Εξωτερικέ έρευνε τι είναι. Είναι έρευνε όπου δεν εμπλέκονται υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή ε, αμοιβόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. πολλές φορές έχουμε και εσωτερική και εξωτερική εμπλοκή. Και το άρθρο 7.4 που μπήκε στον κανονισμό του, της Όλαφ για να ε, είναι δυνατός ο συνδυασμός των δύο διαδικασιών. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπλησιάζει πάρα πολύ τους κανόνες για την εσωτερική και εξωτερική έρευνα στο άρθρο 11.3 εγώ επειδή το θεωρώ σημαντικό, το τόνισα ξανά και ε, θεωρώ ότι δεν δικαιολογείται αυτή η διαφορά, η ε, διαφοροποίηση σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε καλούς κανόνες ε, για όλες τις έρευνες και αυτό είναι και πιο εύκολο για τους ενδιαφερομένους να καταλάβουν ποιοι κανόνες διέπουν την έρευνα που γίνεται της βάρος και ποια δικαιώματα έχουν οικονομικά και πώς μπορούν να τα ζητήσουν. Με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιπλέκεται ε, το νομικό πλαίσιο και το κανονιστικό που ρυθμίζει τις έρευνες της Όλαφ. Δεν είναι μόνο η απάτη, ε, είναι ε, και κάποιες ε, ατασταλίες και παρατυπίες που ε, είναι εκτός της απάτης, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ένα κατόφλι από το οποίο και πάνω επεμβαίνει. Ό,τι βρίσκεται από εκεί και κάτω θα πρέπει να το κάνει όλα. Άρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ερευνά συμπληρωματικά. Και αυτή η διάκριση εσωτερικής και εξωτερικής έρευνας θα ερχόταν να προσθεθεί και να επιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και μετά από τις διάφορες συζητήσεις και τις διελκυστίδες τελικά ε, αποφάσισα να μειώσουμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε αυτή την περιπλοκότητα. Τα δικονομικά δικαιώματα λοιπόν του διαφερομένου με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Έχω κάνει και τροπολογίες και το είχα πει. Δηλαδή να ξεκαθαριστεί το καθεστώς του γραφείου του Ευρωβουλευτού. Αυτό είναι μια παλιά απονεμένη ιστορία. Και πολύ ε, αργά στις διάφορες έρευνες και διαδικασίες χρειάστηκε να επέμβουμε και δεν μπορούσαν ε, να το ε, χρησιμοποιήσουν για λόγους διαδικαστικούς και αυτό είναι μια πραγματική τομή για τον ενδιαφερόμενο. Έγραψα ότι θα πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβαση στο τελικό ε, κείμενο της έκθεσης όλα. Μετά υπήρχε μια πρόταση το 2014 που ακόμα δεν την έχουμε επεξεργαστεί. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει έναν ελεγκτή που ε, θα πρέπει να ελέγχει τις καταγγελίες και τα παράπονα. Ε, ανέτρεξα σε αυτόν τον ελεγκτή και τον έχω προσθέσει στην Εποπτική Επιτροπή είναι η μόνη περίπτωση που η Εποπτική Επιτροπή μπορεί να ελέγχει τρέχουσες διαδικασίες. Κατά τα άλλα περιορίζεται μόνο στις ε, έρευνες που έχουν κλείσει. Επίσης δημιούργησα ε, μια δυνατότητα για τους ενδιαφερομένους να μπορούν να προσβάλλουν και να ακυρώνεται η έκθεση της Όλαφ. Και ποιοι κανόνες ισχύουν ε, υπό τη μορφή κατεξοδότηση πράξεων. Ε, θα θυμάται η συνάδελφος Ινές Αγιάλα, είχατε ζητήσει να γραφτεί ε, ε, στον κανονισμό τον ίδιο στο κείμενο. Εκεί λίγο αγωνιστήκαμε σκληρά, αλλά χάσαμε στο, απέναντι στο Συμβούλιο. θα πρέπει να κωδικοποιήσουμε τι μπορεί να γίνει και πώς θα γίνει. Συμφωνώ ότι θα πρέπει από το, αυτό το εγχειρίδιο να γίνει κατεξουδότηση πράξη. Για να δούμε αν μπορούμε να το υπερψηφίσουμε ή να το καταψηφίσουμε. Αλλά δεν χρειάζεται εμεί να ανακατευτούμε στην ουσία με αυτόν τον τρόπο. Άλλε τροπολογίε. Κατάργηση των IPPs που είναι προτεραιότητε προτεραιότητες Είδαμε και στην Όλαφ ε, ότι είναι και γραφειοκρατικό και βαραίνει τις Ε, η Εποπτική Επιτροπή ε, ε, αφορά διάφορα άρθρα 15, 6α. Επίσης για τις συστάσεις ε, του Γενικού Διευθυντού και πώς δίνουν συνέχεια τα κράτη-μέλη ή τα όργανα. Εδώ λέει μετά από 12 μήνες θα πρέπει το αρμόδιο όργανο το συζητάει με την Εποπτική Επιτροπή. Όχι, μετά από ένα εννέα μήνο προτείνω και σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και τις δικαστικές που τρέχουν στα κράτη-μέλη, επίσης προσθέτω κάποια αιτήματα, καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δημιουργία μια διαδικασία απόλυσης ε, του Γενικού Διευθυντή ε, ε, της Όλαφ. Κύριε Ήταλα, μην το πάρετε προσωπικά, αλλά τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ σκόπιμο και λογικό ε, να υπάρχει διαδικασία. 13 ε, ε, Δευτέρου προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών στις 2 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις, 14, στις 4 Μαρτίου και τον Απρίλιο θα πάει στην Ολομέλεια. Αυτά. Και διάθεσή σα για να σα εξηγήσω οτιδήποτε μπορεί να σα ενδιαφέρει και να έχετε ερωτήσει. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα το λόγο τώρα αν θέλουν ή σκιώδη. Ο κύριο Κόν, παρακαλώ. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εμπεριστατωμένη έκθεση. Ε, ιδιαίτερα μακροσκελής μάλιστα. Αυτό που ε, θέλω να πω είναι ότι σε μεγάλο βαθμό στηρίζω την έκθεση. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι <clears throat> τα μέτρα τα οποία προτείνονται <clears throat> έχουμε ε, πρέπει να βελτιώσουμε τις δικονομικές εγγύησεις, ε, κυρίως όσον αφορά τη συνεργασία με τον ε, εισαγγελέα. Και πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία επικαλύψεις όσον αφορά τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Όλαφ. Ένα θέμα είναι εκείνο το οποίο λιγάκι με προβληματίζει και αυτό το θέμα αφορά στον κανονισμό τι ακριβώς θα γίνει με κράτη-μέλη τα οποία δεν ε, συμμετέχουν, δεν έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς μπορούμε να βρούμε σαφείς κανόνες έτσι ώστε η όλη διαδικασία να έχει νόημα και να είναι και νομικά κατοχυρωμένη. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, και εδώ είναι σημαντικό να υπάρχουν και τα απαραίτητα μέτρα συνέχειας. Όσον αφορά τώρα την εποπτική αρμοδιότητα της αρμόδιας επιτροπής, εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς καλά. Αυτή η εποπτική επιτροπή, ο ελεγκτής, αν δεν μπορεί να καταθέσει δεσμευτικές προτάσεις, τότε σε αμφίσιμες περιπτώσεις ε, πώς ακριβώς θα μας βοηθήσει. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε από αυτού και επίση ε, να δούμε κατά πόσον οι αρμοδιότητες της, ε, του επόπτη, του ελεγκτή πρέπει να διευρυνθούν ή όχι. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Όπως επίσης και τα γραφικά των Ευρωβουλευτών να αφαιρεθούν από τις αρμοδιότητες της Όλαφ. Εγώ δεν συμμετείχα ε, στην τελευταία αναθεώρηση και θα μιλήσω με την κυρία Γιάλα Σάντα για να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το θέμα λογικά. Πέρα από αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στον ε, ΦΠΑ ο οποίο ε, εμπίπτει στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπογραμμίζω αυτό και θέλω να προτείνω κατά την αξιολόγηση του κανονισμού για την Όλαφ όλο αυτό το θέμα πρέπει να το προσαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά από πέντε χρόνια να ελέγξουμε τις εξελίξεις και βεβαίως αναλόγω ε, να ε, άρουμε και τα προβλήματα που ενδεχομένω θα έχουν εντωμεταξύ προκύψει. Κατά τα άλλα υπάρχουν κάποιες ε, διατυπώσεις επί των οποίων πρέπει να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι προσβλέπω στην περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία. Αυτό που είπατε για την αξιολόγηση είναι πάρα πολύ καλό και λυπάμαι που το ξέχασα. Ο κύριο Στάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή ιδιαίτερα η σύνδεση Όλαφ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διευκρινίζεται αυτή. Η δική σας έκθεση, κυρία Γκρέσλε, επίσης με ικανοποιεί, την βρίσκω αρκετά καλή. Τρία πράγματα βρίσκω ιδιαίτερα θετικά. Πρώτον και κυριότερον, οι περισσότερες προτάσεις που κατετίθεται έχουν εμπνευστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την Επιτροπή της Όλαφ ή από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και εμείς ως πράσινοι το υποστηρίζουμε αυτό πάρα πολύ. Δεύτερον, αυτό που λέτε ε, να καταργηθεί η διάκριση που γίνεται ανάμεσα στις εξωτερικές και τις εσωτερικές έρευνες θα πρέπει να ε, εγγυηθούμε ότι η εξουσία και η δύναμη που έχει η Όλαφ θα εξακολουθεί να ισχύει και για εσωτερικές έρευνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτο στοιχείο. Αυτή η υποχρέωση που αντικαθιστά τη δυνατότητα που υπήρχε στο παρελθόν να αρχίζει έρευνα σε περίπτωση απάτης και διαφθοράς η Όλαφ. Δηλαδή τώρα είναι υποχρεωμένη η Όλαφ, δεν δύναται απλώς και το στηρίζουμε απολύτως αυτό ως πράσινη. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που μας προβληματίζουν και έχουμε ένα ερωτηματικό εκεί. Έχω την αίσθηση ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στο παρελθόν στο εσωτερικό της Όλαφ και βγάζουμε διδάγματα από αυτά, αλλά και ο σημερινός ε, γενικός διευθυντής και η επόμενη ε, είναι κάπως εκτεθειμένοι. Δεν ξέρω, μήπως να το διατυπώσουμε διαφορετικά, θα φέρουμε κάποια τροπολογία σχετική. Άλλο πρόβλημα. Το θέμα των ευρωβουλευτών και των διαπιστευμένων βοηθών τους. Ε, να εξαιρείται αυτό από, από την Όλαφ και να εμπίπτει στις ποινικέ ε, διώξεις και έρευνες που κάνουν τα κράτη-μέλη. Εκεί έχουμε προβλήματα εμείς οι πράσινοι. Ε, υπάρχει το καθεστώς ε, των βουλευτών, το οποίο σίγουρα δεν αμφισβητούμε εμείς, αλλά να αποκλείουμε την Όλαφ όταν πάει κάτι στραβά και φταίει ο Ευρωβουλευτής ή ο διαπιστευμένος βοηθός του να εξαιρείται, νομίζω αυτό το παρατραβάει. Και θα, να περιμένετε τροπολογία μας ε, σχετικά. Αυτά σύντομα από πλευρά των Πρασίνων για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Νόβακοφ, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ε, σκιώδης συνέχεια. Ο συνάδελφο Νόβακοφ. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, είναι σωστή. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια τα κράτη-μέλη και οι πολίτες των κρατών μελών έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχει ανάγκη υπηρεσία, η οποία θα έχει την δυνατότητα ε, να ε, απομονώσει παρατυπίες και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με αυτές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ευρύτερη αυτή η η υπηρεσία και η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας αυτής μπορεί βεβαίως να βελτιωθεί σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε έχουμε ξανασυζητήσει τα θέματα αυτά. Τώρα όμως διαπιστώνω ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Όλαφ ε, θα μπορούσε να βρει μια ακόμα καλύτερη μορφή προστασίας των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις προτάσεις του, πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο σε βάθος. Αλλά ε, όταν μιλάμε για τα καθημερινά ας πούμε ε, στοιχεία με τα οποία ε, ασχολείται η Όλαφ μπορούμε σαφώς να υποστηρίξουμε την πρόταση. Πρέπει να βρεθούν όμως και άλλοι τρόποι παρέμβασης ε, της υπηρεσίας στις διάφορες διαδικασίες διερεύνησης κακής χρήσης ή κατάχρησης πόρων εντός των ευρωπαϊκών χωρών. Ε, και θα πρέπει να έχει δυνατότητα παραπομπής προς το δικαστήριο γιατί μερικές φορές η έρευνα δείχνει κάποια αποτελέσματα ωστόσο τα κράτη-μέλη δεν ακολουθούν τις συστάσεις της Όλαφ και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσει κανείς στους πολίτες. Επομένως εγώ υποστηρίζω όλες τις προσπάθειες ενδυνάμωσης των αρμοδιοτήτων της Όλαφ και οπωσδήποτε την διεύρυνση των ικανοτήτων της και την αύξηση της αποτελεσματικότητας σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, πιστεύω ότι η Όλαφ μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά και βεβαίως περιμένω την ώρα των τροπολογιών και της ψηφοφορίας και ευελπιστώ ότι θα, ολοκληρώσει, θα ολοκληρωθεί η εργασία σε τούτη τη θητεία γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, θα απαντήσω στη συνέχεια διάφορα σχόλια. Δεν βλέπω Αλλού παρακαλώ το γύριο γενικό Ιταλ. Α, συγγνώμη, ναι, σας είναι δυνατόν, δεν σε είδα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την εργασία την οποία έχετε κάνει. Ευελπιστούμε ότι ε, θα ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε πριν από το τέλος της ε, θητείας, ε, τουλάχιστον να έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, για να είμαι ειλικρινής, που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση εργασίας. Άλλωστε θα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και μαζί και μπορώ να συμφωνήσω και με όλα αυτά που είπε ο κύριος Κον προηγουμένως και ε, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μία ας πούμε μεταβατική περίοδο ε, ε, ανάμεσα στην εισαγγελία και την ας το πούμε νέα Όλαφ είναι σωστό να γίνει τώρα η αναθεώρηση έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Συμφωνώ και με τον κύριο Στάες ότι ο κανονισμός έρχεται σε μία στιγμή ιδιαίτερη που έχουμε ξεπεράσει και την ε, συγκρουσιακή κατά κάποιο τρόπο σχέση με την ε, Όλαφ και νομίζω ότι σωστό είναι να προβληματιστούμε ε, εκ νέου όσον αφορά τις σχέσεις της Όλαφ και της Επιτροπής Επιτήρησης έτσι ώστε η συνεργασία να είναι ακριβώς πιο συνεργατική και λιγότερο συγκρουσιακή. Ε, γιατί και η Όλαφ και η Εποπτική Επιτροπή έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και βεβαίως εμείς πρέπει να επαγρυπνούμε έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητη απολύτως ε, η Όλαφ. Επίσης, εμείς από την αρχή είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη ε, και όλα τα δικαιώματα, των, τα δικονομικά δικαιώματα των ελεγχομένων ε, και επομένως και οι ερευνητές ας πούμε της ε, Όλαφ ε, θα πρέπει να μην ξεπερνούν τα όρια τα οποία τους έχουν δοθεί και τούτη τη στιγμή είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε τον προβληματισμό μας και την ε, σκέψη μας, πάντα ε, λαμβάνοντας υπόψη την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Όλαφ και της Εποπτικής της Επιτροπής. Γιατί σε αυτήν την μεταβατική περίοδο υπάρχουν κάποιες φαιές ζώνες ε, και ε, δεν ξέρουμε, πρέπει να ξεκαθαριστεί η Όλαφ ποιες αποφάσεις μπορεί να πάρει, σε ποιες κινήσεις μπορεί να προχωρήσει, η Εποπτική Επιτροπή το ίδιο. Ε, και πάντα και σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε εάν θέλουμε η Εποπτική Επιτροπή ε, να λειτουργήσει σωστά, αντί να δημιουργήσουμε νέες επιτροπές και αν θέλουμε πραγματικά αυτή η Εποπτική Επιτροπή να μπορεί να παίξει αυτόν τον διαιτητικό ρόλο με την έννοια ότι να μπορεί να ελέγχει ότι η Όλαφ κάνει αυτό που πρέπει ε, και πληρεί τα καθήκοντά της ε, και λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και προωθεί τις αποφάσεις αυτές, τότε θα πρέπει να δούμε ξανά την εντολή Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο παραπάνω, γιατί ένα πράγμα είναι ε, η εντολή που μερικές φορές είναι πιο περίπλοκη, άλλες φορές πιο απλή και ε, ε, ε, άλλο είναι να λέμε ότι η Εποπτική Επιτροπή με την Όλαφ θα πρέπει να συνεργαστούν και να συμβιώσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο και άλλο πράγμα είναι να ξεκαθαρίζουμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβει η υπόψη της η Όλαφ, ποια είναι τα όρια και τα περιθώρια εντός των οποίων πρέπει και οφείλει να λειτουργήσει. ¿no? Por lo ε, θα πρέπει βεβαίως να ενισχυθεί η εντολή και να προβλέψουμε και κάποιες δυνατές ε, ε, δυνατότητες που θα έχει για το μέλλον, αυτές οι διατητικές ας πούμε ικανότητες που ανέφερα προηγουμένως. Η Εποπτική Επιτροπή θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο ε, ρόλο και να μην, έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, κάποιες ε, αρχές, κάποιες προσφυγές κτλ. Σίγουρα πρέπει να εργαστούμε ε, έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, να διευκρινιστούν οι διαδικασίες να είναι ξεκάθαρες γιατί διαφορετικά ε, θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες και αντιπαραθέσεις στο μέλλον. Και αντιπαραθέσεις λέω και μεταξύ ε, των ιδίων των θεσμικών μας οργάνων. Όσον αφορά τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, εγώ νομίζω ότι τα δικονομικά δικαιώματα και εγγυήσει, ε, ε θα πρέπει να εγγυώνται. Ε, ίσως ε, κάποια κατεξουσιοδότηση ε, πράξη που θα καλύπτει, θα παρέχει την απαραίτητη νομική κάλυψη. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο τι μπορεί κανείς να κάνει και τι όχι, γιατί ξέρετε ότι οι διαδικασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επομένως ε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ε, τα οικονομικά δικαιώματα των ελεγχομένων γίνονται σεβαστά για να μην δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Οι διαδικασίες σαφώς θα πρέπει να είναι δημοκρατικές ε, γιατί εμείς είμαστε κοινοβούλιο και δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι μερικές φορές τα κριτήρια ε, ε, είναι πολύ σωστά και πρέπει να ακολουθούνται και άλλες φορές όχι και τόσο. Πάντως θα συνεργαστούμε με τους υπολείπους συναδέλφους έτσι ώστε να βελτιώσουμε το κείμενο το οποίο αποτελεί ήδη μια πολύ καλή βάση και πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλο κανένα. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Ιταλά, έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, Είμαι ευγνώμων που μου δίνετε τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία ε, Γκρέσλερ, την εισηγήτρια, για την τόσο ολοκληρωμένη έκθεση πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ως Γενικός Διευθυντής ε, της ε, Όλαφ, ε, χαίρομαι για τον προβληματισμό σας όσον αφορά ε, την ε, Όλαφ και την ειλικρινή σας διάθεση ε, για βελτίωση της Όλαφ μέσω της εκθέσεώς σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν τον, έναν κοινό στόχο, την καλύτερη προστασία των συμφερόντων της ενώσεως και των πολιτών της. Και επομένως και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ελέγχου ε, και επίσης δυνατότητα πρόσβασης ας πούμε σε τραπεζικούς λογαριασμούς ε, και εντολή της Όλαφ ε, για δυνατότητα διερεύνησης των στοιχείων αυτών. Υπάρχουν πολλά πιεστικά ζητήματα όσον αφορά πρόσβαση της Όλαφ σε πληροφορίες. Ε, έχετε υποβάλει περαιτέρω τροπολογίες έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών, ας πούμε, ε, όπως θέματα ε, του προληπτικού ελέγχου, της κατοχής προσωπικών ιδιαίτερων εργαλείων και εξοπλισμών κλπ. Ε, ίσως η κατάργηση της διαφοροποίησης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών να είναι κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό και από εκεί θα προκύψουν πολλές τροπολογίες. Θα πρέπει να ε, μελετηθούν πολύ προσεκτικά όλα τα στοιχεία αυτά, να μελετηθεί και ο αντίκτυπός τους, αλλά και η προθεσμία έγκρισης της πρότασης. Επίσης σημειώνω ότι ε, στην έκθεση ε, ε, ζητάτε περισσότερα ενισχυμένα δικονομικά δικαιώματα. Ας πούμε, προτείνει το σχέδιο γνωμοδότησης ότι η Όλαφ με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τα δικονομικά δικαιώματα έτσι όπως αυτά αναφέρονται στην εντολή της Εισαγγελίας. Θα πρέπει επίσης να ξαναδούμε τη λογική της πρότασης της ε, Κομισιόν. Δεν αντιτίθεται ε, στην βασική αρχή των συστάσεων της Όλαφ που δεν είναι δεσμευτικές ε, και που η Όλαφ μπορεί να κάνει διοικητικέ έρευνες και όχι έρευνες σχετικά με ποινικέ διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα καλά ισορροπημένο πακέτο το οποίο ε, θα αφορά και τις δυνατότητες διενέργειας ερευνών από την Όλαφ και την δυνατότητα αποδοχής κάποιων στοιχείων ως αποδεικτικών ε, τεκμηρίων. Τέλος καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται ε, σε αδέκαστη και αντικειμενική καλή συνεργασία. Κατανοώ και συμμερίζομαι τον προβληματισμό που εκφράζεται στην έκθεση για, την, ε, για τις σχέσεις με την Όλφα. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της σχέσης δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εσαΐ εμπλοκής της μίας υπηρεσίας ή ε, του ενός οργάνου από το άλλο έτσι ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις ε, ακινησίας. Αυτό που προσπαθεί η Κομισιόν ε, είναι να συζητηθεί ε, το θέμα αυτό και με τούτη τη θητεία του Κοινοβουλίου και με την επόμενη ε, ε, θητεία που θα ξεκινήσει σε λίγο. Προσδοκούμε λοιπόν σε καλή μελλοντική συνεργασία και με την εισαγγελία έτσι ώστε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καλύτερα να διασφαλιστούν. Η Κομισιόν προσπαθεί ε, να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του κανονισμού Όλαφ μέχρι το 2020 όταν θα αρχίσει δηλαδή να είναι λειτουργική και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επομένως ενθαρρύνω την Επιτροπή σας ε, να μην το λησμονεί αυτό και επομένως να εστιαστεί στο τι μπορεί να γίνει μα βράχει πρόθεσμα έτσι ώστε ε, η Όλαφ και η αποστολή της για προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, να ευοδοθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την ειλικρίνεια. γνωριζόμαστε εδώ και καιρό και τα προβλήματα που έχει Όλαφ εξακολουθούμε να τα μετακυλίουμε από χρόνο σε χρόνο. Τώρα τι θα κάνουμε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία ή θα τα λύσουμε. Προσπαθήσαμε να λύσουμε κάποια πράγματα, καταφέραμε να επιβάλλουμε και ορισμένα άλλα. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα και πρέπει να σας το πω. Και το πρόβλημα αυτό ποιο είναι και είναι πάρα πολύ δυσεπίλητο. Και κάθε τροπολογία έχει δύο όψεις και θα πρέπει πάντα να δισταθμίζουμε αυτά τα πράγματα, τι θέλουμε. Και ε, ε, ε, σε ποιο κύμα θα σερβάρουμε πρώτα. Και πάντα είναι τα διλήμματα έντονα. Ε, και δεν υπάρχει μια βασιλική οδός, αλλά πρέπει να σταθμίσεις και να επιλέξεις. Λοιπόν, ακούω τώρα και βλέπω ότι κάνει το Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο είναι έτοιμο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι πριν το Συμβούλιο, πριν καταλήξει καν σε κοινή θέση. Και τι κάνει το Συμβούλιο. Τα σβήνει αυτά από την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, εμείς τα προσθέτουμε. Και αυτή είναι μια θαυμάσια βάση. Αν δεν καταφέρουμε τίποτα να, να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, δεν θα συμφωνήσει και το Συμβούλιο. Και για κάθε πρόοδο θα πρέπει να σκαρφιζόμαστε διάφορα τεχνάσματα για να διαπραγματευόμαστε με τα κράτη-μέλη. Δεν ήταν ευχάριστο την περασμένη φορά. Εγώ είμαι προθυμή να προχωρήσω γρήγορα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί τι συμβιβασμού θα προτείνει ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε εμεί, σε αυτό που θέλει το Συμβούλιο. Αλλά το το, ο συμβιβασμός δεν είναι να βγει κάτι να περάσει από το θέμα αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω κάτι για την ασυλία. Γιατί είναι σημαντικό για πολλούς συναδέλφους. Αν λέει το κοινοβούλιο ότι έχει υποβάλει ε, ταξιδιωτικά έξοδο βουλευτής και το βρίσκει ύποπτο, Μπορεί Όλαφ να το ε, ερευνήσει, αλλά όχι να μπουκάρει στο γραφείο του Ευρωβουλευτή. Εγώ ε, τα ειστήρια μου τα δίνω στη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Έχει πρόσβαση η Όλαφ εκεί και μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να ε, γίνεται φασαρία πολιτική στα γραφεία των βουλευτών. Εφόσον αφορά κάτι το γραφείο ενός Ευρωβουλευτή, θα πρέπει προηγουμένως να ε, γίνει σε εθνικό επίπεδο η άρση της ασυλίας και να κάνει τη δουλειά της η Όλαφ. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική και στα κράτη-μέλη. Αλλιώς είναι αδιανόητο να, κάνει έφοδο η Όλαφ στα γραφεία μας. Ξέρω ότι δίστανται απόψεις, θα το ψηφίσουμε. Για μας στη Γερμανία είναι αδιανόητο Γίνονται διοικητικέ έρευνες, αλλά αυτή η ιστορία με την απάτη ε, και ε, ε, τα ταξιδιωτικά έξοδα, της δαπάνη, τα οδηπορικά, τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά, όλα αυτά τα δίνουμε στη διοίκηση και τι δουλειά έχει το γραφείο του βουλευτού. Από εκεί και πέρα. Για τον έλεγχο. Και τον έλεγκτη του δώσαμε το δικαίωμα ήδη αυτή τη στιγμή έχει κάνει τον έλεγχό του να επιβάλλει κάποια πράγματα στο Γενικό Διευθυντή. Γι' αυτό είναι αλλαγή στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθήσα να αντιγράψω κάποια πράγματα που μου είχαν υποδείξει άλλοι. Με πιάνει και ένα δέος, είναι πάρα πολύ βαριά αυτή η δουλειά. Και δεν ήθελα να μπω σταύρο σε ιαλοπολείο και να τα κάνω όλα λίπα. Αλλά με βάση την εμπειρία μου της τελευταίας πενταετίας ή επταετίας, πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί έχω δει ότι δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ είναι πανίσχυρος. Ε, σε όλη τη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, είναι εκείνος που κινεί όλα τα νήματα. Είναι μεγάλη εξουσία του. Κανένας άλλος γενικός διευθυντής δεν έχει τόση εξουσία όσο ο γενικός διευθυντής Όλαφ, ουδής. Και νομίζω ότι είναι ευφυές να προσθέσουμε και κάτι και να πούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον ε, ένας με τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία που να μην είναι πάντα αντιπαράθεση με τριβές και καυγάδες και θετική. Προσπάθησα λοιπόν να κάνω μια ανεξάρτητη έτσι, αρχή, ε, γιατί αν δεν το γράψουμε στον κανονισμό δεν πρόκειται να επιβληθεί ποτέ. Ε, οι εμπειρίε του παρελθόντος μόνο κακές ήταν. Προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα, δεν ξέρω αν προκαλούμε τώρα καινούργια, θα δείξει. Πάντως ευκαιρία το θεωρώ. Και επίση ε, θέλω πραγματικά να υποστηρίξω την κατεξουσιοδότηση πράξη. Η Όλαφ είναι καλύτερη μοίρα από οποιοδήποτε άλλο όργανο. Ότι θα πρέπει να κωδικοποιούμε τις διαδικασίες, ιδιαίτερα μια τέτοια υπερεθνική διαδικασία. Ε, είστε οι μόνοι που μπορείτε να πείτε κάτι. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να κωδικοποιήσει τις διαδικασίες, αυτή είναι η Όλαφ. Και νομίζω ότι πραγματικά χρειάζεται να το κάνουμε. Γιατί αυτό είναι και το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκοποίησης εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουμε σωστές διαδικασίες. Μου είπε κάποιος πρόσφατα τις προάλλες ότι ε, με την Όλαφ θα πέσετε σε ένα νομικό μεσαίωνα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε ένα νομικό μεσαίωνα ε, για να λύνουμε προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει από μόνο του κάθε κράτος μέλος. Χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και δυνατότητα προσφυγής, να ε, ε, έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να προσφεύγει με αποτελεσματικότητα. Δηλαδή όταν κάνει κάποιος προσφυγή για αποζημίωση να μην περιμένει 15 χρόνια στο Βέλγιο ας πούμε. Θυμάμαι με ένα επίτροπο για ένα δάνειο που δεν έχει δικαιωθεί. Τι να πει και ο απλο πολιτη άμα χρειάζεται τόσο βαριέ και χρονοβορε διαδικασιε Σημείωσα αυτό που είπε η Νέσα Γιάλα για τι φαιέ ζώνε. Είναι τόσο πολλέ αυτέ οι γκρίζε ζώνε. Να τι φωτίσουμε λίγο. Ξέρω ότι σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί αυτό και όλα θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει καλύτερα, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να κάνω. Τόσο μπορώ. Ο κύριος και πάλι, παρακαλώ. Ναι, θέλω λίγο να επανέλθω όμως παρόλα αυτά. Στην αρμοδιότητα που πρέπει ή δεν πρέπει να έχει όλα και την εξουσία να κάνει έρευνες διοικητικές, δεν λέω. Για ευρωβουλευτές ή διαπιστευμένους βοηθούς τους. Για μένα είναι αδιανόητο να κάνουν έφοδο στα γραφεία των βουλευτών. Στο παρελθόν το έχουμε ζήσει αυτό. Και ήταν ξεκάθαρο ότι κάποιοι βουλευτές απασχολούσαν κάποιους υποτίθεται διαπιστευμένους βοηθούς οι οποίοι δούλευαν για το κόμμα. Κάτι ακροδεξιοί τύποι μου έρχονται στο μυαλό. Αυτό είναι σαφής παραβίαση των κανόνων και του καθεστώτος του βουλευτού και του ε, διαπιστευμένου βοηθού αν κάνει διοικητική έρευνα η Όλαφ, γιατί έχουν έρθει καταγγελίες, καλώς κάνει. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάει να ψάξει μερικά πράγματα και στο γραφείο του βουλευτή. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να μην συνάδει ε, με τα ήθη και τα έθιμα στα κράτη-μέλη που προστατεύονται οι βουλευτές με κάποιο διαφορετικό τρόπο, αλλά από την άλλη αυτός μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος να γίνει μια κανονική έρευνα σωστή. Αυτό γιατί να το αποκλείσουμε. Και οι ίδιοι οι ερευνητέ τη Όλαφ ε, μπορούν να αποφασίσουν κατά την κρίση του αν χρειάζεται να πάνε σε ένα γραφείο ευρωβουλευτή. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, πάντα θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση και συμφωνία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα. Προφανώ δεν θα μπουκάρουν στο Κοινοβούλιο, κάνουν έφοδο, γεια σα, ήρθαμε και φέρτε εδώ τα έγγραφα. Υπάρχει και ένα σωστό τρόπο συντακτικό και συντεταγμένο για να τα ε, ερευνήσει αυτά. Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, με τον Γενικό Γραμματέα και ίσως και με τη φυσική του παρουσία. Υπάρχει τρόπος να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα σωστά. Τώρα διαφωνούμε από ό,τι φαίνεται, δίστανται απόψει. Αλλά σας λέω και πώς το βλέπω εγώ. Πολύ συχνά, λέει ο κύριος ε, Τσιτσόφσκι, έχουμε την αίσθηση ότι εδώ βλέπουμε ταινία τρόμου ε, και η Όλαφ μπαίνει ξαφνικά φορώντας μαύρα ρούχα στο γραφείο των βουλευτών στο κοινοβούλιο, κραδένοντας το όπλο της και λέγοντας εγώ είμαι η Όλαφ και τα λοιπά. Γιατί, γιατί να πρέπει η Όλαφ να μπορεί να μπει στα γραφεία των βουλευτών. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ από την, πλευρά μου, ναι, έχει δυνατότητα η Όλαφ να και έχει δικαιοδοσία και έχει και την εξουσία να κάνει έρευνες εάν πιστεύει ότι ε, εγώ έχω κάνει κάποια απάτη. Αλλά το, ζήτημα εδώ δεν είναι να αμφισβητήσουμε αυτό το δικαίωμα της Όλαφ, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κάνει την έρευνα η Όλαφ. Θα υποβληθούν όλα τα στοιχεία και τα λοιπά χωρίς κανένα πρόβλημα φυσικά. Αλλά δεν πρέπει να γίνει εδώ ταινία western. Jenom pro to samotné vyšetřování Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν, με, δεν αμφισβητώ τη δυνατότητα έρευνας, αμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διεξαχθεί η έρευνα αυτή. Δεν είναι θα μπει όλα αυτά καουμπόις, ας πούμε, και να τα κάνει όλα λίμπα. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Όλαφ να μπορεί να μπαίνει στα γραφεία των βουλευτών. Είναι τόσο απλό. Ίσως ε, ε, δεν καταλαβαίνω από τεχνικής απόψεως πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα. Also, nehmen wir mal an, ναι, λοιπόν, α υποθέσουμε ότι έχω πάρει ένα έγγραφο από κάποιον που το κρίνω ότι είναι σοβαρό έγγραφο, σημαντικό. Και με αυτό μπορώ να δουλέψω. Και μετά προσπαθεί η Όλαφ ε, να πάρει και αυτή αυτό το έγγραφο και έρχεται στο γραφείο μου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η δουλειά των Ευρωβουλευτών επηρεάζεται πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία. Περί αυτού πρόκειται οι έρευνε τη ε, Όλαφ κατά μίας ε, πολιτικής ομάδας η οποία τους ε, ε, βοηθούς τους έβαλε να δουλεύουν για το κόμμα, αυτή η είσοδο έγινε απρόσκοπτα στα γραφεία αυτής της πολιτικής ομάδας. Αλλά παλιότερα τι συνέβαινε. Συνέβαινε ότι μπορούσε να μπει η Όλαφ μόνο εάν είχε τη συνένεση του Ευρωβουλευτή. Και νομίζω στην τελευταία αυτή έρευνα πήραν ένα hard disk, το σκληρό δίσκο των υπολογιστών. Εκεί όμω σε αυτό το σκληρό δίσκο υπάρχουν πληροφορίε και για άλλου ευρωβουλευτέ. Άρα η δουλειά ενό ευρωβουλευτή αφορά και του άλλου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προστατευόμαστε. Ε, πρέπει να προστατεύουμε ακόμα και εκείνου ε, των οποίων δεν συμμερίζομαι την πολιτική τοποθέτηση. Ε, όσον αφορά του βοηθού, ε, εκεί μπορεί όλα να κάνει ό,τι θέλει. Να δει τι συμβάσει, να δει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει. Ε, τώρα το θέμα του ε, να είναι παρόντες ή κατά πόσον οι ε, βοηθοί είναι παρόντες στα γραφεία, κατά πόσον δηλαδή πράγματι δουλεύουν ή όχι, αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Και αυτό μπορεί όμως κανείς να το ελέγξει ε, χωρίς να μπει απαραίτητα στο γραφείο. Μπορεί κανείς να το ελέγξει παραδείγματος χάρη ελέγχοντας ε, τα μπάτζι τις ε, κάρτες αυτές για να μπει κανείς στο κτίριο. Και επίσης και με άλλους τρόπους. Έτσι έγινε με αυτή την πολιτική ομάδα που σας λέω. Είδανε ότι αυτοί οι βοηθοί δεν ερχόντουσαν να δουλέψουν εδώ, αλλά δούλευαν μάλιστα σε τελείως διαφορετική πόλη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τροπολογιών, τι να σας πω. από καθαρά ευρωπαϊκή σκοπιά, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό που είπε η Όλαφ, ότι αγοράστηκαν κάποιες τροπολογίες, ε, δεν ξέρω ε, κατά πόσο. αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Όλαφ. Ε, αυτά εμπίπτουν προφανώς στην εθνική δικαιοδοσία. Τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Τέλο πάντων, εγώ ε, προτίθεμαι να προστατεύσω τη δουλειά των ευρωβουλευτών, αλλά επίση ε, προτίθεμαι να κυνηγήσω και αυτούς που είναι μικροαπατεώνες. Τώρα, ε, τα θέματα των ε, δαπανών, ταξιδίου κτλ. Νομίζω ότι αυτά η όλα μπορεί να τα ελέγξει γιατί έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα στο Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω ότι όσον αφορά το να μπαίνουν στα γραφεία μα, εκεί διακυβεύονται πάρα πολλά. Το να μπορούμε να δουλέψουμε. Ε, και εγώ εκλήθην ως μάρτυρας για κάποια έκθεση και τους έγραψα μια πολύ ευγενική επιστολή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα παρουσιαστώ. Δεν θέλω δηλαδή κατά κάποιον τρόπο να αλλάξουν τα κριτήρια με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Θεωρώ ότι το όλο θέμα είναι σοβαρό και ως εκ τούτου η διοίκηση του Κοινοβουλίου τότε ε, κατέθεσε τις ε, τροπολογίες, εγώ τις πήρα, τις ανέσυρα και νομίζω ότι ήταν καλό να παραμείνουν. Το Συμβούλιο αρνήθηκε την τελευταία φορά, ενδέχεται να αρνηθεί και αυτή τη φορά, αλλά εγώ θέλω να συζητήσω μαζί τους ε, και να τους πω, συγγνώμη, τι τίμημα ε, πρέπει να καταβάλουμε. Δεν εννοώ προφανώς κάθε τίμημα, είναι σαφέ, αλλά νομίζω ότι κατά τη δική μας την άποψη ε, θα έπρεπε και εξάλλου, αυτό είναι και το κείμενο δίκαιο, δηλαδή υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και έχει κάπως εκτονωθεί η κατάσταση, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του Γενικού Διευθυντή, κατά πόσον οι διαδικασίες που ήδη τρέχουν, κατά πόσον τα βρίσκεται όλα αυτά σωστά ή όχι. Γιατί πρέπει να σας πω το εξή. Ένα σκληρό δίσκο από τους δικούς μας υπολογιστές δεν θέλω να φτάσει σε άλλα χέρια γιατί εκεί υπάρχουν στοιχεία και για άλλους, για πολλούς. Κύριε Γενική Διευθυντά, παρακαλώ έχετε το λόγο. Βεβαίως ε, αυτό το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δηλαδή το ε, πώς ακριβώς θέλετε εσείς να αντιμετωπίσετε και να χειριστείτε το θέμα. Αλλά εγώ μέχρι τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, εντάξει συνέβη κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά τα τελευταία χρόνια η Όλαφ ποτέ δεν έχει βάλει στα γραφεία. Εμείς καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν σε εμά να συζητήσουμε μαζί τους, αλλά άρχισα νομίζω, άρχισαν να γίνονται συζητήσεις ε, με το Γενικό Γραμματέα, με τον κύριο Βέλε. Έχω αρχίσει να συζητάω μαζί του σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Όλαφ και το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η πεμπτουσία του θέματος. Δεν ξέρω αν δηλαδή θέλετε να έχετε αυτή την τροποποίηση του κανονισμού, γιατί αν το διαβάζω σωστά, Ίσως να μην είναι απόλυτα σαφές ότι όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τα γραφεία και αυτή είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. γιατί αν δεν εγκριθούν κάποια θέματα, ποτέ δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε τα κράτη-μέλη, ακόμα και αν έχουμε αποχρώσεις ενδείξεις για απάτη ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Αν λοιπόν θέλετε να υπάρξει αυτή η αλλαγή, πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι εδώ πραγματικά εννοούμε τα γραφεία, φυσικά γραφεία για τα έγγραφα και για όλα τα σύναφη. Δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος και βεβαίως ίσως να είναι χρήσιμο για τη συζήτηση σας με το Συμβούλιο το να είναι το Κοινοβούλιο ο μόνος χώρος όπου να μπορούμε να εισέλθουμε και να ε, ανακρίνουμε ανθρώπους αν υπάρχουν ε, σαφείς ενδείξεις για απάτη. Αλλά σας λέω, είναι καθαρά πολιτικό το θέμα ε, και νομίζω θα πρέπει να είναι σαφής η τροπολογίες. Και τώρα που τα διαβάζω δεν είμαι και σίγουρος ότι όλα αυτά είναι απόλυτα σαφή. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Θα το δουλέψουμε λιγάκι για να δούμε τι ακριβώς εννοείτε κι εσείς. Πραγματικά όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα και αυτά τα οποία κάνουμε είναι πρωτοποριακά. Ε, μέχρι τώρα δεν έχει πράξει τίποτα από αυτού και γι' αυτό το λόγο ε, πρέπει να συζητήσουμε με τους ε, ενδιαφερόμενους, να είμαστε βέβαια απόλυτα σαφείς. Και τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, έχω τη βούληση να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια. Εχθές έγινε μια συζήτηση ανάμεσα στους συνεργάτες μου και την Όλαφ. Και στις ε, προτάσεις που καταθέσαμε ε, ρωτάμε μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Συγγελία αν δεχτεί ερώτηση από την ε, Όλαφ. Υπάρχει κάποια, κάποιος χρονικός περιορισμός. νομίζω κάτι υπάρχει. Γίνεται λόγος για κάποιες ημέρες, αλλά νομίζω η Όλαφ χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Εγώ τη διάρκεια την τροπολογία, αλλά με πάση περιπτώσει μάλλον πρέπει να το ξαναβάλω, γιατί επ' αυτού θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Θα καταθέσω σχετική τροπολογία. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε συνάντηση των σκιωδών, να μου πούν οι συγγιστέ, πότε τους ε, βολεύει και ε, θα προσπαθήσουμε το όλο θέμα να το διεκπαιρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη συζήτηση και να σας πω ήδη τώρα ότι αυτά τα οποία θα προκύψουν πραγματικά είναι πολύ σημαντικά. Να έχουμε μια πιο αποτελεσματική Όλαφ, καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη δουλειά της Όλαφ. Αυτό πραγματικά μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε τελικά να μην κερδίζουν οι απαταιώνες, αλλά το κράτος δικαίου. Βεβαίως το κράτος δικαίου θα πρέπει και αυτό να είναι δεσμευμένο σε κάποιους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ για την όλη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντά που ήρθατε και να είστε σίγουρος δεν θα χαθούμε. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 7. για την αποστολή αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στη Σλοβακία. Ο συνάδελφος Βόν ήταν επικεφαλής, γιατί εγώ ε, πηγαίνοντας στο Κόσιτσα αποκλείστηκα στη Βαρσοβία. Εκεί κατέληξα. Ε, σας ευχαριστώ όλους και όσοι συμμετείχαν εκεί. Ήταν πολύ σημαντική. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Βόν για να μας παρουσιάσει την αποστολή αυτή, την έκθεσή της. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, λέει ο κύριος Βόχαν, όλους αυτούς που πήγαν ε, στην Σλοβακία και συμμετείχαν σε αυτήν την συνεδρίαση πρέπει να σας πω ότι ε, συνήθως αυτές οι αποστολές ε, είναι, και, είναι πολύ ενδιαφέρουσες και τούτη εδώ στη Σλοβακία δεν αποτέλεσε, ε, δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Πρέπει δεν να σας πω ότι είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και από τον τύπο. Είχαμε πολλούς διερμηνείς, συγγνώμη, πολλούς δημοσιογράφους ε, και διότι η διερευνητική αποστολή έγινε και μετά από την δολοφονία ε, του, των ε, δημοσιογράφων και μάλιστα να σας πω ότι είχαμε και πολλούς γεωργούς με πανό, μάλιστα είδα ένα πανό που έλεγε παρακαλώ βοηθήστε μας κυρία Γκρέσλερ πραγματικά περιμένουν πολλά από μας. Είχαμε τρεις μέρες ε, ε, διάρκεια της αποστολής, αλλά πολύ εντατικές αυτές ε, οι μέρες. Μιλήσαμε, συναντήσαμε πολλούς γεωργούς, τρεις ομάδες γεωργών ε, που ήθελαν ε, χωριστές ε, συναντήσεις. Τα μηνύματα πάντως ήταν περίπου ίδια από όλες τις ομάδες των γεωργών και τα παράπονα ήταν τα ίδια. Τα κύρια παράπονα των γεωργών ήταν ότι δεν μπορούν να ζητήσουν γεωργικές επιδοτήσεις γιατί αυτές ταυτόχρονα τις ζητούν για τις ίδιες γέες μεγάλες εταιρείες οι οποίες ε, φαίνονται να είναι δικαιούχες ε, των άμεσων πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, μας μετέφεραν εκφοβισμό των γεωργών, φυσικές απειλές. Μας έδειξαν τέτοιες φωτογραφίες. Μας είπαν, μάλιστα, ένας νέος γεωργός, ο οποίος με πολύ συγκινησιακό τρόπο μας είπε ότι θέλει να μείνει σε αυτή τη δουλειά, θέλει να είναι γεωργός, αλλά δεν μπορεί να μείνει ως ε, γεωργός λόγω των προβλημάτων ε, που σχετίζονται με, ε, με την αδυναμία του να πάρει αυτές τις άμεσες επιδοτήσεις. Το πρόβλημα λοιπόν, το κύριο πρόβλημα ήταν η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για επιδότηση. Πέρα και γύρω από, το πρόβλημα αυτό υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα εκφοβισμού των ε, γεωργών. Συνδεδεμένο δε με αυτό είναι και το θέμα της ε, ε, ειρήνης, του ειρηνικού περιβάλλοντος στην Ήπεθρο. Γιατί λόγω ακριβώς των πολλών συμβάντων και περιπτώσεων εκφοβισμού και φυσικής βίας οι γεωργοί φοβούνται, οι χωρικοί φοβούνται υπάρχουν δε από ό,τι μας είπαν διασυνδέσεις των μεγάλων εταιριών πολύ συχνά και με κυβερνητικά στελέχη ε, και επομένως ε, τις περισσότερες, ε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βρίσκει κανείς το δίκιο του και επίσης μας κατήγγυλαν ότι ακόμα και σε περίπτωση απατών δεν βρίσκεται άκρη και δεν δικάζονται, δεν καταδικάζονται τελικά οι υπεύθυνοι της απάτης όταν αυτοί είναι μεγάλες εταιρείες ή μεγάλοι γεωκτήμονες και και ε, ε, ε, σε πολλές περιπτώσεις μας κατήγγυλαν ότι οι υπηρεσίες γεωργικών πληρωμών, αυτές οι APAs, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και πολλές φορές μας είπαν ότι οι υπηρεσίες, η υπηρεσία γεωργικών πληρωμών ακόμα και ενώπιον των δικαστηρίων δεν, δεν αλλάζει τακτική. Ένα άλλο σημείο ήταν το εξής. Ε, σε περίπτωση διαφωνίας ε, όσον αφορά τον δικαιούχο της ε, επιδότησης συστήνεται στον δικαιούχο μικρό γεωργό να πάει στα δικαστήρια αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ περιπλεγμένα γεωργοί εντωμεταξύ δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους δεν μπορούν γιατί δεν έχουν πάρει καμία επιδότηση και μοιραία οδηγούνται στην πτώχευση. Αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά στοιχεία ε, της συζήτησης και με την Υπηρεσία Γεωργικών ε, Πληρωμών που φαίνεται ότι ε, θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι την δικαιοδοσία να ελέγξουν την υπόθεση, να δουν ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος της άμεσης πληρωμής έτσι ώστε να μην στραγγαλίζονται οι μικροί γεωργοί. Επίσης ε, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, ένας ε, κυβερνητικός ε, νόμος που πέρασε τελευταία και που δεν δίνει την δυνατότητα στους μικρούς γεωργούς να εκθέσουν τα ε, ζητήματά τους ε, έτσι ώστε να βρουν τα δίκια τους. Ε, μιλήσαμε επίσης και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, μιλήσαμε και με εισαγγελείς, συναντήσαμε εισαγγελείς και είδαμε τι μπορεί να γίνει με τις ε, ε, διώξεις ε, όσον αφορά αυτές τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις καταβολής των επιδοτήσεων στην υπηρεσία γεωργικών πληρωμών είδαμε μεγάλο δισταγμό όσον αφορά την απάντηση ε, των ε, ερωτήσεών μας. Είδαμε πάρα πολύ αμυντική στάση ε, του επικεφαλής, ο οποίος δεν είχε διάθεση να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Επίσης, συζητήσαμε με τον, συναντήσαμε τον Υπουργό Γεωργίας. Μας είπε ότι δεν ε, καταλάβαινε γιατί βρισκόμαστε ε, στην ε, Σλοβακία και αναγκαστήκαμε να εξηγήσουμε στην Υπουργό τι έννοια έχουν οι διερευνητικές επιστολές, συγγνώμη, αποστολές του Κοινοβουλίου και ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία μας έχουν υποβληθεί. Στο τέλος είχαμε συνέντευξη τύπου Είχαμε πολλούς ε, ε, δημοσιογράφους και στο τέλος ε, κάναμε κάποιες συστάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πάντα κάποιες συστάσεις στο τέλος των ε, το, των αποστολών αυτών ε, και έχουν, θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοι να δουν και τις, ε, τις συστάσεις που κάναμε. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και τους ε, ε, Σλοβάκους ε, γεωργούς να ακουστεί η φωνή τους. Θα πρέπει επίσης και το Υπουργείο να τίνει ευήκονους έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά την μη καταβολή των επιδομάτων, το πρόβλημα των διπλοετήσεων πληρωμών και επιδοτήσεων και επίσης ε, θα πρέπει η υπηρεσία γεωργικών πληρωμών να κατανοήσει ότι θα πρέπει καλύτερα να λειτουργεί και ότι θα πρέπει η ίδια να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να λύνονται τα προβλήματα αυτά. Συστήσαμε επίσης να ε, ξαναδεί και η κυβέρνηση την ε, νομοθεσία για την αναθεώρηση της χρήσης γης ε, ξέρετε, στην Σλοβακία υπάρχουν πάρα πολλοί μικρές ε, ιδιοκτησίες, 20-30 ε, τετραγωνικά πόδια και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Επίσης συστήσαμε να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το θέμα των μισθωμένων γεών και ίσως ε, βάσει ενός κτηματολογίου θα πρέπει να ε, δίνεται απόδειξη της, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της γης ε, πριν ετηθεί κάποιος επιδόματος. Επίσης είπαμε περαιτέρω μέτρα να ληφθούν έτσι ώστε να επιβληθεί σωστά ο νόμος στην Σλοβακία. Μπορούν να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορούν μπορεί να βελτιωθεί η ε, λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών που σχετίζονται με όλη αυτή την κατάσταση. Αυτές είναι οι συστάσεις. Ε, στείλαμε ε, την έκθεση στους συναδέλφους οι οποίοι έστειλαν με τη σειρά τους πίσω κάποια, κάποιες παρατηρήσεις και βεβαίως εάν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να συζητήσουν περαιτέρω είμαι στη διάθεσή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Τεχόφσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Τέρεκ Βον ε, για την ε, ηγεσία της ε, αποστολής. Ήταν πολύ σκληρή η επιστολή. Μας λείψατε πρόεδρε, χάσατε τη πτήση σας. Αλλά ο Ντέρεκ επάξια σας εκπροσώπευσε ήταν ε, όσο γινόταν πιο ουδέτερος και πιο αμερόληπτος καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής. Προσπάθησε να ακούσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, σε όλα τα προβλήματα και θέλω να τον ευχαριστήσω. Ε, περιέγραψε κάποια από τα πράγματα που βρήκαμε εκεί. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι λίγο διαφορετικό, αν μου επιτρέπετε. Εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ ε, για τη γεωργική πολιτική και την διαφθορά στη Σλοβακία. Εδώ και χρόνια. Είμαι από τους λίγους εδώ ε, μεταξύ ημών που καταλαβαίνω τα σλοβακικά και έχω ίσως κάπως καλύτερη αίσθηση από τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας. Ήταν η τρίτη αποστολή που πήγε φέτος στη Σλοβακία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ σοβαρά τα προβλήματα διαφθοράς στη Σλοβακία. Ο Ντέρεκ είπε ότι είχαμε αποδείξεις εκφοβισμού και βίας κατά των γεωργών και κατά οποιοδήποτε καταγγέλει, καταδεικνύει ε, αδικία και απάτη τους κρατάνε τις ε, πληρωμές, τους αποσύρουν τις επιδοτήσεις. Θα πρέπει να το προσέξει πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράδειγμα, έχουμε αποδείξεις ενονικά ότι κάποιος έσπηρε σιτάρι στο χωράφι του και έρχεται κάποιος και του κλέβει τη σοδιά. Και πάει και του ζητάει το λόγο ο πρώτος αγρότης, μα τι κάνεις, πήγες και μου θέρισες το σιτάρι και τον συλλαμβάνει η αστυνομία. Το πρώτο, αυτό που είχε σπείρει το σιτάρι. Έχουμε και βίντεο και στοιχεία και ό,τι άλλο θέλετε, αλλά η αστυνομία διαφορεί. Άλλο πρόβλημα που έχουμε εμεί στην τσεχική δημοκρατία. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν μπορούν να πάρουν ευρωπαϊκέ επιδοτήσει. Έχουμε πρόγραμμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και τελικά επειδή στο τέλος της περίοδου δεν μπορέσαμε να κάνουμε το διαγωνισμό και να απορροφηθούν τα κονδύλια, συμπεριλάβαμε και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες σιγά σιγά άρχισαν να αγοράζουν ό,τι υπήρχε στην αγορά από γη. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει και στη Σλοβακία. Μετά από αυτή την αποστολή λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε ότι πήραμε δεκάδες email και επανειλημμένα έχω συναντηθεί ε, με γεωργούς, με καταγγέλλοντες δημοσίου συμφέροντος, αστυνομικούς, νυν και πρώι που μου έδειξαν διάφορα πράγματα která není prošetřena. Předražených zakázek. Zak για διαφθορά, για διάφορα εγκλήματα διαφθοράς, δικήματα που μένουν αδιερεύνητα, για διάφορες για διάφορους διαγωνισμούς στο Κομάρνο, για νέες μηχανές τα οποία μηχανήματα, τα καινούργια που παίρνουν, είναι σε χειρότερη μοίρα μετά από ένα χρόνο από ότι ε, άλλα τα παλιά της 20 ετίας. Όλα αυτά λοιπόν που είδαμε στη Σλοβακία θα πρέπει να έχουν και κάποια συνέχεια, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ε, ταυτόχρονα, όπως είπε και ο Ντέρεκ, εξακριβώσαμε ότι ήμασταν ανεπιθύμητοι εκεί ως αντιπροσωπεία. Και πρώτη φορά ήμουν εγώ σε μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου μας μίλησαν και μας φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο όπως μας φέρθηκαν στη Σλοβακία. Είναι πραγματικά έσχος αυτό. Για να θυμηθούμε το πλαίσιο όμω. Σκότωσαν ένα δημοσιογράφο και τη μνηστή του. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται να διερευνηθεί αυτό. Ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπόλ επίση. Διότι η Ευρωπόλ βοήθησε ε, να διερευνηθεί ε, όλη αυτή η υπόθεση και να συλληφθούν οι, ε, οι πέτοι. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω, για να ενισχύσουμε την έκθεσή μας, να γράψουμε διάφορα πράγματα. Πρώτον, η γεωργική μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητα, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Σήμερα τι ισχύει. Έχεις 100 τετραγωνικά τα οποία έχουν 14 ιδιοκτητε. Χαιρετίσματα. Αυτό ευνοεί πολύ την απάτη. Υπάρχει μια τεράστια καχυποψία των αγροτών απέναντι στη δημόσια διοίκηση. Και θα πρέπει να τους πούμε οπωσδήποτε και συστηματικά να ζητάμε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να βγάλουν τα αποθυμένα τους και να προσπαθήσουν να προχωρήσουν και να βρουν μια λύση. Η σημερινή σχέση που έχουν, γι' αυτό το περιγράφει ο Υπουργό Γεωργίας και ε, Γεωργών δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα διάλογο και αυτό δεν μπορεί παρά να επί, ε, την κατάσταση. Επίση, οι υπηρεσίε που ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι συχνά ε, διεφθαρμένες, έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας και ζητούν και εμείς οι ίδιοι. Και η τέταρτο αυτό που ζητάω τώρα, θα πρέπει να κοιτάει τι γίνεται με τις αγορές που κάνουν για επενδυτικούς λόγους ε, σε διάφορα γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες, ε, θεριζόλνιστικές μηχανές κτλ. Ε, το σλοβακικό σύστημα προμηθειών πρέπει να εξεταστεί. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, ένα τρακτέρ που κάνει 100.000 ε, στην Αυστρία να κάνει 180.000 στη Σλοβακία. Και τα έχουμε δει αυτά με στοιχεία αποδεδειγμένα. Να δούμε τι γίνεται με τα γεωργικά ταμεία. Αγοράζουν κάμερες, ξέρω εγώ, που υποτίθεται θα πρέπει να είναι για την πυροπροστασία. Ε, δεν δουλεύουν οι κάμερες και είναι και υπερτιμημένες. Ε, Πολλέ φορές πολλαπλασιασμένη η τιμή του. Επίσης να ενισχυθούν οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις για κάποιου αγρότες που θέλουν να φημώσουν. Γιατί μας τα λένε όλα αυτά οι αγρότες. Και μάλιστα όσοι μας μίλησαν την άλλη μέρα τους στείλανε επιθεώρηση ε, στην εκμετάλλευση. Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν τέτα μυρίζει. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση, αλλά εγώ δεν την καταλαβαίνω ή περιπτώσεις αγροτών που κατέδειξαν προβλήματα και τους ήρθε η επιθεώρηση το Δεκέμβριο. Και δεν ολοκληρώθηκε κιόλα για να μην κλείσει ο χρόνος ε, και να μην πάρουν τις επιδοτήσεις και να περάσει το διάστημα και να είναι 3,5 χρόνια και όχι τρία. Όπως και ο νεαρός αγρότης τον οποίο σε εσύ, ε, Ντέρεκ δίνουν γεωργικές επιδοτήσεις για χώρους στάθμευσης, ξέρω εγώ, ή για ε, ασφάλτους στρωμένους δρόμους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το ξαναδούμε το σύστημα αυτό γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι μικρομεσαίοι κλήροι δεν παίρνουν καθόλου επιδοτήσεις ενώ τα περισσότερα, τα, μάλλον όλα τα λεφτά τα παίρνουν οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Και αυτά ε, είναι πολύ λίγοι άνθρωποι. Η κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ. Έχουν υποθεί ήδη πάρα πολλά. Ο Ντέρεκ Βόρν ήταν θαυμάσιος πρόεδρος στην αντιπροσωπεία και φυσικά μας έλειψε η πρόεδρος, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Η έκθεση του Ντέρεκ ε, είναι πάρα πολύ φιλική. Αν την είχα γράψει εγώ θα τα είχα πει πολύ πιο έξω από τα δόντια. Συνοψίζω λέγοντας ότι δεν ήμασταν καθόλου ευπρόσδεκτοι βγήκαν και μας είπαν καλά γιατί μας ξανακουβαληθήκατε. Τώρα προχθές φύγανε οι προηγούμενοι. Τι κάνετε πάλι εσείς εδώ. Και προσπάθησαν να μας ε, συντρίψουν ε, με ε, οι αρμόδιοι υπάλληλοι από τη ε, μάζα και τον όγκο των στοιχείων που μας φέρανε. Από κάθε τμήμα ήταν ένα εκεί με ένα βουνό χαρτιά. Δεν το καταφέρανε αυτό. Ε, υπάρχει το γραφείο συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά τι κάνει αυτός εκεί ο επικεφαλής. Υπάρχει κανένα σύνδεσμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με ε, την κυβέρνηση. Γιατί αυτός ε, είχε μια στάση του στυλ κάνω ό,τι μου λέει η κυβέρνηση και κατά τα άλλα βοήθεια γιατί με κυνηγάνε. Ε, ήταν πολύ φιλικός ο άνθρωπος, δεν λέω, και ευγενικό, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με σύνδεση του Κοινοβουλίου με τον κόσμο εκεί επιτόπου. Ε, συμφωνώ και με τον Τόμας Δεχόφσκι. Υπήρχε σύγκρουση πάντα από τη μια οι αγρότες με τα αιτήματά τους ε, που είναι σίγουρα δικαιολογημένα και από την άλλη ε, οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Είχαμε παρόν και ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου που κατά τα άλλα δεν άνοιξε το στόμα του, δεν πήρε ποτέ το λόγο και αυτό με εξέπληξε. Δεν ξέρω, μπορεί έτσι να συνηθίζεται ή μπορεί εκ των υστέρων να προκύψει κάτι που να μας πει τι, τι σκεφτόταν αυτή η κυρία από το ελεγκτικό συνέδριο. Πάντως μας είπανε ότι οι απαντήσεις για τους αγρότες που δεν έχουν τα χωράφια τους δεν έρχονται από ε, το Υπουργείο Γεωργίας αλλά από κάποιους εξωτερικούς τους οποίους έχει ανατεθεί αυτό. Στην Deloitte συγκεκριμένα το έχουν αναθέσει και υπάρχει και ένας πρώην επάλληλος της Deloitte που δουλεύει τώρα στο Υπουργείο Γεωργίας και είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε. Και ρωτήσαμε... Καλά, πριν ε, βγάζατε 11.000 ευρώ καθαρά στην Deloitte και τώρα πήγατε στο Υπουργείο για να βγάζετε 2.500 και είπε ότι καλά, η καταπληκτική εμπειρία που ζω τώρα στο Υπουργείο δεν πληρώνεται με τίποτα καλά προσπάθησαν πραγματικά να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, ε, να φτιάξουν ένα ε, χωριό τύπου χωριού ποτέ, Ποτέμκιν, να μας παρουσιάσουν την ωραία εικόνα. Ε, πραγματικά εγώ θα έλεγα την έκθεσή μας να την γράψουμε με τρόπο πολύ πιο οξύ και με ύφος πολύ πιο οξύ για να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Δηλαδή, να το ζήσουμε αυτό, να το δούμε αυτό και να τα αφήσουμε χωρίς συνέπειες δεν επιτρέπεται. Και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που είναι καθαρός συνεισφορέα και τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε, δεν επιτρέπεται να τα αφήνουμε να υπάρχουν. Γιατί έτσι γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αναξιόπιστη τι θα κάνουμε τώρα, θα κλείσουμε το στόμα μας και θα τα συγκαλύψουμε, αλλά αν πούμε κάτι να το πούμε ε, πηγόντως και να έχουμε και το θάρρος να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να βγάλουμε και τα συμπεράσματα και τις συνέπειες. Ο συνάδελφος Στέφανετς. like Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία ε, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την δύσκολη αλλά τόσο ε, σημαντική αποστολή κυρίως για τους μικρούς γεωργούς της Σλοβακίας. Ένα σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω. Υπόθηκε και προηγουμένως ε, το μήνυμα από την κυβέρνηση ακόμα και από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό, την Υπουργό εμ, Γεωργίας ήταν γιατί δεν κατανοούσαν τον λόγο ύπαρξης αυτής της αποστολής, γιατί γινόταν αυτή η αποστολή. Η Λουμπίτσα Βόσκορα ε, κατηγορήθηκε από την ε, από την ε, αστυνομία για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κυρία ε, δέχτηκε πάρα πολλές, ε, μάλλον ήταν υπεύθυνη για πάρα πολλές ε, καταγγελίες που έγιναν από μικρούς γεωργούς. Άρα το μήνυμα που δόθηκε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και για αυτό που είπε ο συνάδελφος Τόμας προηγουμένως, δηλαδή πολλοί γεωργοί που συναντήθηκαν μαζί μας έχουν μπει στο στόχαστρο της ε, διοίκησης ε, που τους στέλνει διαρκώς ε, επιθεωρήσεις και μάλιστα στείλανε αμέσως επιθεωρήσεις μετά από την αποστολή μας και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν είναι εγκληματική ενέργεια η συνάντηση με την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ απλώς προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους όσον αφορά την καταβολή των επιδομάτων. Ε, είναι πολλοί οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν τη γη τους, αλλά τελικά, ενώ είναι δικαιούχοι, δεν παίρνουν ε, τις ε, γεωργικές επιδοτήσεις. 75% των επιδοτήσεων πηγαίνουν στις τσέπες των μεγάλων γεωργών. ενώ στην, στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο οι μικροί γεωργοί, ενώ είναι η πλειοψηφία, διαρκώς η θέση τους χειροτερεύει και δεν παίρνουν τελικά τα επιδόματα, ενώ έχουν κάθε δικαίωμα να τα πάρουν. Ε, είναι γεγονός ότι δεν είναι πολύ σαφές βάσει της νομοθεσίας ποιος είναι ο δικαιούχος ε, των ε, επιδοτήσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να αναμορφωθεί ο σλοβακικός νόμος να ε, ε, φαίνεται ότι το καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς και άρα μόνο αυτός που είναι ιδιοκτήτης ή αυτός που έχει μισθώσει γη ε, και την καλλιεργή είναι δικαιούχος να λάβει τα, γεωργικά, τις γεωργικές επιδοτήσεις. θα πρέπει το ξεκαθάρισμα να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Σλοβακίας και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ντέρεκ ότι δηλαδή χρήζει απολύτως αναμόρφωσης ο γεωργική νομοθεσία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και η Σλοβακική κυβέρνηση. Επίσης, πολλές είναι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ε, υποβάλει συγκεκριμένα παράπονα και καταγγελίες. Κρίμα είναι να μην αναφερθούμε σε, αυτές, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, οι συναντήσεις αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν ε, ε, τροφή για σκέψη και ενδεχομένως για ε, να σκύψει πάνω στα θέματα αυτά η εισαγγελία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει κάτι να γίνει. Ελπίζω ότι δεν θα τελειώσει αυτή η κατάσταση με αυτή την έκθεση και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στη Σλοβακία γιατί πρέπει να γίνει αυτό για να γίνουν και ουσιαστικές αλλαγέ. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ έχω ζητήσει να μιλήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ήμουνα στην ε, Βαρσοβία και δυστυχώς ε, έχασα την ανταπόκριση. Μου κλείσανε την πόρτα στο πρόσωπο, κατά πρόσωπο. Ε, δυσάρεστη εμπειρία αυτή για μένα, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό ήταν να είμαι και εγώ παρούσα και πόσο σημαντικό ήταν να τα δει κανεί αυτά επί τόπου να τα βιώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα λέτε έτσι όλα τόσο ανάγλυφα. Έχω κάποιε ερωτήσει για να δούμε πού ακριβώ ε, είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι μια, ένα ερώτημα προ την κυρία Μπόχμαν από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Με ενδιαφέρει τα συμπεράσματα, τα συμπεράσματά σα γιατί ήσασταν παρούσα. Και θα ήθελα να σα το δείξω λιγάκι αυτό. Αυτό που βλέπετε το πορτοκαλί είναι τα ποσά, οι ενισχύσει στο των 100.000 ευρώ και Και βλέπετε ότι 13% ε, μετά πάνω από 100.000 ευρώ έχουν φτάσει στο 70%. Δηλαδή μιλάμε για το πιο άδικο σύστημα που υπάρχει εντωμεταξύ στην Ευρώπη. Ο αριθμό εκείνων που παίρνουν 100.000 ευρώ είναι το 7% όλων των δικαιούχων. Το 7% παίρνουν το 70% των κονδύλιων. Συγγνώμη, αυτό ε, προφανές κάτι δεν πάει καλά. Και τώρα μία ερώτηση προς την κυρία Μπόρχμαν. Ε, τι πρέπει να αλλάξουμε στο ενωσιακό δίκαιο. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα και τι ακριβώς μάθατε από όλα αυτά. Τι κάνετε εντωμεταξύ και τι συμβουλεύετε εμάς. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς κάθε τρεις μήνες θα το βάζουμε το θέμα στη μερίσια διάταξη. Θα το κάνουμε αυτό, θα επιμείνουμε όπως και με την Ουγγαρία και με όλες τις άλλες χώρες οποίες ε, ε, βέβαια ε, επιβαρύνουν τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ σκεφτόμουν τι πρέπει να πω έχοντας ακούσει τους μετέχοντες. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μάλλον που με δεχθήκατε στην αντιπροσωπεία που μετέβει επί τόπου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι και πρέπει να σας πω ότι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπαν οι αντιπροσωπείες, οι νέοι γεωργοί, αλλά όλοι οι γεωργοί θα έλεγα, η ΜΚΟ και πολλοί άλλοι που μίλησαν για την κατάσταση στη Σλοβακία. Και ε, τα συμπεράσματα που εξήγα εγώ από την επίσκεψη αυτή είναι ότι πραγματικά πρέπει να υπάρξει κάποια παρακολούθηση στην ε, Σλοβακία. Και μάλιστα πιστεύω ότι το σχέδιο της ε, έκθεσης είναι απόλυτα σαφές ε, γιατί ξεκαθαρίζει ποια είναι τα προβλήματα και χαίρομαι που επίσης ξεκαθαρίζει ότι η αντιπροσωπεία δεν μπόρεσε επιτόπου να επιβεβαιώσει τις ε, αιτιάσεις ή την έκταση αν θέλετε των αιτιάσεων. Εκεί πρέπει να υπάρξει κάποια συνέχεια. Και επίσης πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά το θέμα. Ελπίζω να μην μπω σε πολύ τεχνικά θέματα, αλλά όσον αφορά καταρχήν τις υποψίες για απάτες. Αυτά τα παρακολουθεί βεβαίως η Όλαφ. Και εμείς από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας παρακολουθούμε τις γεωργικές ενισχύσει. Η Όλαφ λοιπόν θα εξετάσει το θέμα των υποψιών για απάτη. Επ' αυτού θέλω να πω ότι, όπως είπα και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ήταν καλό η Επιτροπή να αποκτήσει αντίγραφα από όλα αυτά, γιατί η αντιπροσωπεία πήρε πάρα πολλά έγγραφα που εγώ δεν τα πήρα, πραγματικά σωρό, τεράστιο σωρό εγγράφων και πρέπει και εμείς κάπως να τα δούμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να το παρακολουθήσουμε το θέμα, ούτε η Όλαφ, ούτε εγώ, αν δεν δούμε τα συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από την επίσκεψη προφανώς και συμπέρανα ότι πρέπει να προκλουθήσουμε και τον ίδιο τον οργανισμό πληρωμών. Και εδώ θέλω να κάνω μία διαφοροποίηση. Εάν έχουμε μία κατάσταση όπου υπάρχει διαφωνία για το ποιος ακριβώς εκμισθώνει τη γη και ποιος ακριβώς καλλιεργεί τη γη, στο βαθμό που μπορούμε να ξέρουμε, ο οργανισμός πληρωμών λέει ε, δεν πληρώνουμε κανένα. Αυτό όμω είναι πρόβλημα για τους ε, μικρούς ε, γεωργούς, αλλά δεν είναι πρόβλημα, αν θέλετε, για τις γεωργικές ενισχύσεις, γιατί προφανώς δεν έχουν καταβληθεί. Τέλος, η απόφαση λαμβάνεται είναι ότι πληρώνεται, καταβάλλεται η ενίσχυση στον πιο μεγάλο γεωργό, γιατί αυτός αντέχει και περιμένει. Προφανώς ε, και θα πρέπει να εξετάσουμε τον οργανισμό πληρωμών και αυτό το κάνουμε εμείς ως Επιτροπή. Και να διαφοροποιήσω λιγάκι και ανάμεσα σε δύο άλλα πράγματα, γιατί ο κύριος Σερτσόφσκι προηγουμένως ανέφερε ότι ε, καταβάλλονται πάρα πολλές ενισχύσεις ε, για τα τρακτέρ. Αυτή είναι η γεωργική εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, όχι απόλυτα, ενδιαφέρεται με τις άμεσες πληρωμές και ε, όσον αφορά αυτές τις ε, άμεσες ε, πληρωμές και εκεί πρέπει να εξεταστεί το θέμα κατά πόσο υπάρχουν απάτες ή όχι. Αλλά πράγματι πρέπει να παρακολουθήσουμε λιγάκι αυτούς τους οργανισμούς πληρωμής. Γιατί αυτοί λένε ότι έχουν μόνο 40 περιπτώσεις που εναπομένουν από το 17 που τελικά ήταν 18. Αλλά σας λέω και πάλι αυτό είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπέτρου και τις ε, δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται οι και συνεχίζονται και τα προγράμματα δράσης ε, για την ε, Σλοβακία. Θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε και ε, θα δούμε αν πρέπει να γίνουν κάποιες δημοσιονομικές διορθώσεις. Δηλαδή, το θέμα των δημόσιων διαγωνισμών δεν είναι καινούριο. Αν υπάρχει απάτη, είναι θέμα της Όλαφ, ε, αλλά και το θέμα είναι ε, να δούμε κατά πόσον λειτουργεί καλά το σύστημα με τους οργανισμούς πληρωμών. Το ελεγκτικό συνέδριο της Σλοβακίας το εξέτασε το θέμα και εμείς μάλιστα το είχαμε κάνει πριν από αυτούς ε, άρα γνωρίζουμε ότι αυτό πράγματι, γιατί έχουμε εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Εμείς στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ελέγχουμε τα συστήματα ελέγχου, κατά πόσο είναι σωστά και όσον αφορά τις απάτες σας λέω αυτά τα ερευνά η Όλαφ. Προφανώς ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Όλαφ για ανταλλαγή πληροφοριών και μόλις ε, μας δώσετε και εσείς τα στοιχεία που πήρατε κατά τη διάρκεια της αποστολής, αυτό θα μας βοηθήσει. Υπάρχει βέβαια και ένα τρίτο θέμα ε, προσπαθήσετε να το πείτε λιγάκι στην έκθεση σας. Είναι θέμα κράτος δικαίου, θέμα μεταρρυθμίσεων ε, γεών. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα εδώ η πίεση πρέπει να σκεφτεί περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο. Τι δηλαδή πρέπει να γίνει αν υπάρχει τέτοιο θέμα για τις ε, μεταρρυθμίσεις, τις εκτάσεις στη γη. Υπάρχει ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, και α, όσον αφορά τα, ε, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είναι πάρα πολύ μικρές όσον αφορά τα οικόπεδα καλλιεργήσιμης γης. Ε, ε, αν είχαν όλοι καταχωρήσει τα συμβόλαια εκμίστοσης, αυτό θα βοηθούσε, γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν ε, κάποια, ε, κάποιο συμβόλαιο εκμετάλλευση και εμφανίζεται ξαφνικά στον οργανισμό πληρωμή κι άλλο ένα με το ίδιο συμβόλαιο για την ίδια γη. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο οργανισμό. Πρέπει το θέμα να διευθετηθεί στο Εθνικό Δικαστήριο. Και υπάρχει και ένα άλλο, ε, νομίζω ότι Εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη τι θα παρακολουθήσει όλα και τι θα ε, δούμε εμείς από πλευράς ε, διαχείρισης ε, και οργανισμών πληρωμών. Σας είπα λοιπόν το τι θα εξετάσουμε ε, εμείς ε, ε, θα παρακολουθήσουμε τις άμεσες πληρωμές στην γεωργική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της υπαίθρου, γιατί εκεί έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης των σλοβακικών αρχών. Α, και κάτι άλλο, όσον αφορά την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων και τον επιμερισμό. Αν δείτε λιγάκι τον επιμερισμό αυτό, θα διαπιστώσετε ότι εκεί γίνεται λόγος για τις πληρωμές που έχουν λάβει η χώρα. Αν είναι μεγάλη γεωργή που έχουν τεράστιες εκτάσεις, αυτοί από το 2010 ε, Προφανώ παίρνουν περισσότερα χρήματα και παίρνουν περισσότερα χρήματα όχι απλά επειδή είναι μεγάλη γεωργή, αλλά διότι έχουν αυτό το facing in των ε, άμεσων ενισχύσεων. Από το 2010 το facing in ε, συνεχίζεται, άρα δηλαδή αν έχει κανείς μεγάλες εκτάσεις και παίρνει ε, περισσότερες ενισχύσεις για ανάλογα με την έκταση των εκταρίων, προφανώς και παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα προοδευτικά. Η Σλοβακία και η Τσεχία είναι οι δύο χώρες με κάποιο περίεργο επιμερισμό, κάπως διαφορετικό από τις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να το δει κανεί κάτω από το γενικότερα πρίσμα μεταρρυθμίσεων των άμεσων ε, ενισχύσεων η Κομισιόν μετά το 2020 θα προσπαθήσει να βάλει ένα ανώτατο όριο στις άμεσες ενισχύσεις, να μην μπορεί δηλαδή να λαμβάνει κανείς ένα τεράστιο ποσό. Ε, να υπάρχει και ε, σταδιακή μείωση ε, στις πληρωμές. Νομίζω ότι το όλο θέμα είναι και λιγάκι πολιτικό όσον αφορά τον, το πώς ακριβώς επιμερίζονται οι άμεσες ενισχύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι εδώ κακά αυτά που ακούμε. Ε, μας ε, ενοχλεί ότι δεν έχουν έρθει ακόμα τα έγγραφα τα οποία επίκυνται και είναι σημαντικό για μας κάθε τρίμηνο ε, να μας στέλνετε μια επιστολή και να μας λέτε τι έχετε κάνει. Θέλουμε και εμείς να παραμείνουμε να το παρακολουθούμε, αλλά και εσείς. Και τώρα ελπίζουμε να μην μας λένε κάθε φορά τα ίδια μετά από τρεις μήνες. Μπορούμε να σας παρακαλέσουμε να μας κάνετε μια τριμηνία έκθεση. Τι συνέχεια δίνεται, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πώς έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα feedback και να το μοιράζουμε σε όλους. Γιατί εγώ έχω ανησυχήσει από τώρα με τις γεωργικές επιδοτήσεις ε, σε κάποια κράτη-μέλη, νέα κράτη-μέλη, όχι παντού, η Πολωνία είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε μια νέα γεωργική αριστοκρατία που δημιουργείται, μια νέα τάξη με ευρωπαϊκά κονδύλια και πολλά και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και χάρη σε αυτά επιρροή. Και αντίστροφα η εθνική πολιτική ζει από αυτό, από την εκδίωξη από τις γέες ε, των ε, ε, μικρών ε, γεωργών. Γιατί δεν υπάρχει ε, καμιά ρύθμιση για αναδασμούς ας πούμε, για νέα διάταξη και γεωργικές μεταρρυθμίσεις. Το ξέρω, δεν φταίτε εσείς. Τώρα γεωργική μεταρρύθμιση, αυτό ακούγεται τρομερό, αλλά αν υπάρξει ένας αναδασμός, μία ρύθμιση για το πώς χρησιμοποιούνται τα χωράφια. Θα μου πείτε και αυτό μπορεί να χρειαστεί 20 χρόνια, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσει. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά κονδυλία. Ο συνάδελφο Στεχόφσκι ξαναζήτησε το λόγο και μετά θα παρακαλούσα εσά, κυρία Μπόρχμα. Στα γερμανικά, ε, ε ο Τάμα Στεχόφσκι, θέλω να απαντήσω σε αυτό που είπατε, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα απαντήσω στα τσεχικά. Ο Ντέρεκ ε, Βον. Ε, ε, μάλλον να πω στον Ντέρεκ, μετά την επίσκεψή μας, ορισμένοι γεωργοί άρχισαν να συνασπίζονται, να συνεταιρίζονται. Άρα δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο καταγερματισμό, όπως λες στο τέλος της εκθεσής σου στις συστάσεις. Από ό,τι φαίνεται, πάνε να δημιουργήσουν ένα, μία ένωση γεωργών ή δύο, εν περιπτώσει, για να μπορούν να αντιδράσουν. Στη συνέχεια. Ε, για 120 περιπτώσεις μάθαμε τι έγινε μετά την δική μας επίσκεψη. Εγώ μπορώ αυτά να τα παριθμίσω και με περιγραφή στα αγγλικά. Και αν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό μπορούμε να το ετοιμάσουμε μέσα σε δύο εβδομάδε και να το υποβάλουμε. Συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που πήραμε κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή μα. Και θα πρέπει να δούμε αν η Όλαφ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια θα τα εξετάσουν όλα αυτά τα περιστατικά. Έχουμε ξεχωρίσει κάποιε περιπτώσει, γιατί δεν θεωρούμε ότι ήταν απάτη ή γιατί τα έγραφα. Ε, δεν ήταν σοβαρά. Αυτά τα έχουμε βγάλει στην άκρη. από την άλλη όμως υπάρχουν τουλάχιστον 60 πάρα πολύ συγκεκριμένε και σαφείς περιπτώσεις που χρειάζεται να ε, τις κοιτάξετε. Και από τα έγγραφα βλέπουμε ότι είχαμε συστηματικές παραβιάσεις ε, σε προκηρύξεις διαγωνισμών, ε, σε χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε αυτές οι πληρωμές είναι άμεσες πληρωμές επενδυτικές κλπ. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Κυρία Μπόρχμαν, θα πάρετε τα έγγραφα λοιπόν εσείς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι έχουμε και εμείς ανθρώπους που ξέρουν σλοβαγικά. Δεν χρειάζεται να είναι στα αγγλικά. Βεβαίως η κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Έχουμε δει και εμείς περιπτώσεις για αιτιάσεις και κατηγορίες ε, ε, ε, απάτης. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ εκεί είναι να το διαβεβάσω στην Όλαφ, γιατί εμείς δεν ερευνούμε απάτες. Κυρία Γκρέσλε, μέχρι εδώ όλα κακά, ε, δεν νομίζω. Λάβετε παρακαλώ υπόψη ότι οι καταγγελίε και οι αιτιάσεις που λάβαμε πέρσι αφορούσαν απάτη και διαφθορά. Αυτό δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας ή των εσωτερικών μας ελεγκτών. Αυτά τα ψάχνει όλα Μπορείτε να ζητάτε εκθέσεις κάθε τρεις μήνες, αλλά όπως σας είπα, μέχρι τώρα αυτές οι καταγγελίες που λάβαμε αφορούσαν την απάτη. Άρα τα διαβιβάσαμε αρμοδίως στην όλα. Τι σας λέω, τι εννοώ και τι βγάζω εγώ από την αποστολή αυτή. Ότι μπορεί να υπάρχουν και τα δύο ταυτόχρονα και οι καταγγελίες για διαφθορά και κάποιες άλλες που πρέπει να δούμε το διαχειριστικό και ελεγκτικό σύστημα των πληρωμών, αν λειτουργεί, αν λειτουργεί. Αυτό κάνω αυτό τον καιρό και σας είπα θα εξακολουθούμε να το εξετάσουμε σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα ξέρουμε τα προβλήματα και τα παρακολουθούμε. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα δράσης, μπορείτε να το δείτε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και πραγμένων για τις άμεσες πληρωμές. Βεβαίως και τα παρακολουθούμε. Δεν είναι ότι έχουμε σταυρό στα χέρια και δεν κάνουμε τίποτα. Και μετά για το κράτος δικαίου υπάρχει ο εισαγγελέα, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει ένα κρατικό ταμείο γεών που από ό,τι έχω καταλάβει ε, κατέχει το 20% των γεών. Τώρα όπως αυτά τα, πια, τα εκμισώνει και τα διαθέτει, ε, δεν μας αφορά. Αυτά μας ξεπερνάνε μας ε, ως Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Δηλαδή ποιος θα μισθώσει ποιο χωράφι, αυτό δεν είναι δική μας υπόθεση. Υπάρχει ένα πολιτικό θέμα που θέλει συνέχεια και πιστεύω ότι και οι συστάσεις στην έκθεσή σας θα ε, αντικατοπτρίζουν αυτά πάρα πολύ ωραία. Και σας παρακαλώ, όταν σας λέω ότι θα το παρακολουθήσουμε και το κοιτάμε. Ε, είναι γεγονός και βοήθησε πάρα πολύ η παρουσία μου εκεί για να καταλάβω ακριβώς ε, ότι δεν είναι ακριβώς θέμα απάτης αμυγός. Πρέπει να δούμε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και θα το κάνουμε. Αυτό σας λέω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Περιμένουμε με χαρά να λαμβάνουμε τις τακτικές σας εκθέσεις. Ο κύριος Βόν για να κλείσει. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν βέβαια στην αντιπροσωπεία και την γραμματεία που μας υποστήριξε, καθώς επίσης ε, και να ευχαριστήσω πολύ ε, και το γραφείο των αξιωματούχο ε, σύνδεση στην Μπρατισλάβα από το γραφείο μας πραγματικά ήταν πολύ υποστηρικτική. κοιτάξτε, ε, όπως καταλάβετε και η ήταν πραγματικά δραστήριο μέλος σε αυτήν την αντιπροσωπεία. Ε, νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι μετέφεραν εδώ την στάση των εκπροσώπων της Σλοβακικής ε, κυβέρνησης και λίγο καταλάβαμε και γιατί αισθάνονται ε, τόσο παραμελημένοι και αγνοημένοι από την κυβέρνηση οι μικροί ε, γεωργοί. Να πούμε πάντως ότι από την ώρα που φύγαμε ε, έχουμε ε, κάποιες εξελίξεις, ας πούμε έχουν αρθεί οι κατηγορίες ε, προ, όσον αφορά το πρόσωπο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Επίσης και η Υπηρεσία Γεωργικών Πληρωμών έχει πλέον έναν εκπρόσωπο ο οποίος μιλάει εξ ονόματός της και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη όσον αφορά τις συστάσεις Ε, ε, πολλοί συνάδελφοι έκαναν ε, συστάσεις. Νομίζω πάντως ότι αυτές οι επιμέρους συστάσεις στην ουσία καλύπτονται από τις συστάσεις που αναφέρουμε εμείς εδώ στην έκθεση της διαρευνητικής αποστολής, κυρίως όσον αφορά το, τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, μικρούς γεωργούς κλπ. Νομίζω ότι όλα αυτά ε, αναφέρονται. Μπορούμε βέβαια να προσαρμόσουμε τις συστάσεις ε, κυρίως όσον αφορά ε, και συμβόλαια χρήσης γης αλλά και όσον αφορά εξοπλισμό, τρακτέρ και τα λοιπά. Ναι, μπορούμε να το ξαναδούμε λίγο, να τα προσθέσουμε συγκεκριμένα αυτά. Επίσης ε, ε, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ε, επιδομάτων φαίνεται να πηγαίνει των επιδοτήσεων, συγγνώμη, φαίνεται να πηγαίνουν, να καταλήγουν τελικά στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων. Ε, επίσης, η εκπρόσωπος ε, της ε, Κομισιόν μας είπε ότι θα υπάρχει κάποιο follow-up και εμείς θέλουμε follow-up, κυρίως όσον αφορά κάποιες πληρωμές, να τις έχετε κατά νου λίγο έτσι ώστε όταν θα βελτιωθούν, να, να, να δούμε δηλαδή αν στο μέλλον θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα. Η συνέχεια, το follow-up οπωσδήποτε είναι χρήσιμο Επίσης ε, να σας πω ότι παρότι εμείς ζητήσαμε κάποια τεκμήρια ε, δεν μας δόθηκαν ε, αυτά. Φαντάζομαι ότι η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει περισσότερα αποδεκτικά στοιχεία γιατί και εμείς από τη δικιά μας πλευρά όσο πιο πολλά τεκμήρια έχουμε τόσο πιο καλά μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Πιστεύω ότι στην ε, γνωμοδότηση και κυρίως στις συστάσεις ε, αναφέρονται πολλά από αυτά τα στοιχεία, αλλά βεβαίως ε, εάν κάποιοι κάποια μέλη της αντιπροσωπείας, κυρία Πρόεδρε, έχουν συγκεκριμένες ιδέες, παρακαλώ να τις υποβάλουν. Ευχαριστώ πολύ. Και για τη δουλειά που έχετε κάνει, δεν θα τελειώσει αυτό το θέμα, σίγουρα θα παραμείνουμε ε, τελειώνω όμως το θέμα στη μέση διάταξη και πέραμε στο 8. Ε, ε, ασχοληθούμε το, με το άρθρο 143 του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό τι κρύβει. Ε, μια τράπεζα δεδομένων που λέγεται EDIS ε, για επιχειρήσεις που βαρύνονται με διαφθορά και απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια τράπεζα δεδομένων που αποκλεί τις εταιρείε αυτές. Είναι δικό μας τέκνο αυτή η Επιτροπή. Ε, επανειλημμένα ε, ε συγκρουστήκαμε, αγωνιστήκαμε, ε, δεχτήκαμε πλήγματα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τελικά διατυπώσαμε έτσι το άρθρο ώστε να μπορούμε να ε, δουλεύουμε καλά και χαίρομαι που προεδρεύει στο πάνελ ε, και ε, το πάνελ το οποίο αποφασίζει ποιες εταιρείε θα εγγραφούν σε αυτή την τράπεζα δεδομένων ο κύριος Πενέρα, πρώην νομικό σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ παρόν παρακαλώ σας για το λόγο για να μας παρουσιάσετε λίγο το θέμα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όντως Πάνε πέντε χρόνια από τότε που έφυγα από το Κοινοβούλιο και τώρα επανέρχομαι ε, ως πρόεδρος αυτού του οργάνου, πάνελ, γκρέμιο μου στα γερμανικά όπως θέλετε, ε, για το σύστημα έντις. Τι είναι αυτό το σύστημα έντις. Αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό. 12 σελίδες είναι από 190 Δηλαδή ένα σημαντικό τμήμα του δημοσιονομικού κανονισμού έχει αφιερωθεί σε αυτό το μηχανισμό και σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Είναι και πολλές αιτιολογικές σκέψεις, έχουμε ένα ιστορικό κανονισμό 15 σελίδο περίπου και όλα αυτά λειτουργούν ελπίζω με τρόπο ικανοποιητικό για σας και για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσω λίγο να το εξηγήσω, είναι κάπως περίπλοκο και θα προσπαθήσω επίσης να μην σας ε, κουράσω πάρα πολύ. Ποια είναι η βελτίωση από το δημοσιονομικό κανονισμό του 2018. Δεν είναι μία, είναι πολλές και σημαντικές. Το κείμενο έχει καταστεί σαφέστερα ευανάγνωστο, έχει περισσότερη ουσία και μας διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή. Γιατί στο παρελθόν είχαμε χρονικούς περιορισμούς ε, για τον ε, οικονομικό έλεγχο δηλαδή ε, και για ε, να ακούσουμε τον ενδιαφερόμενο, τον αντιδικό ή όπως θέλετε πείτε το. Ε, έχει ε, περισσότερο χρόνο και να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενδιαφερόμενος και εμείς να ασχοληθούμε με τον έλεγχο. Έχουμε δύο είδους αρμοδιότητες. Μία εσωτερική αρμοδιότητα από την 1η Πρώτου του 2019 έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τις εσωτερικές ατασταλίες Έχουμε αυτή την ευχάρι... Είμαστε στην ευχάριστη θέση, αν μπορώ να το πω έτσι. Για εκείνου που εκτελούν τον προπολογισμό. Είναι μια κεντρική αρμοδιότητα, διοργανική. Ευτυχώ ακόμα δεν έχει αποτανθεί κανεί σε εμά για αυτό το θέμα. Βέβαια είναι λίγε εβδομάδε μόνο που έχουν περάσει. Πάντω είναι θετικά όλα αυτά γιατί εξασφαλίζουν μια ε, συνέχεια εσωτερική. Νομίζω αυτό το λέει το άρθρο 97. Έχουμε όμω και εξωτερικέ αρμοδιότητε, σε αυτέ θέλω να αναφερθώ, που αφορούν ε, πρόσωπα φυσικά και νομικά ε, που ε, λαμβάνουν ε, κατόπιν συμβάσεως χρήματα, τα οποία διαχειρίζονται και ενδεχομένω πρέπει να διωχθούν. Δύο είναι οι περιπτώσεις όπου παίρνουν κοινοτικά κονδύλια άνθρωποι όχι και τόσο είναι εκείνοι που πτωχεύουν, που βέβαια μπορεί να μην φταίνε οι άνθρωποι, για εκείνοι που έχουν ζητήματα με την εφορία ή με την κοινωνική ασφάλιση, τις κοινωνικές εισφορές. Όταν κάποιος ε, διατάκτης έρχεται αντιμέτωπος με τέτοια πρόσωπα, τα αποκλεί. Προς το παρόν έτσι συμβαίνει, μπορούμε να το συζητήσουμε θέλετε γιατί είναι πολλές επιφυλάξεις. Μετά, μπαίνουμε τώρα στην ουσία. Υπάρχουν θέματα και άλλα που είναι αρμόδιο το πάνελ μας σε περιπτώσεις όπου είναι του οργανωμένου εγκλήματος, ε, ε, ε, κακουργήματα, απάτη, διαφθορά, σύμφωνα με την οδηγία προδιετίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, εκείνοι που απασχολούν παιδιά, τρομοκράτες κτλ. Αυτά παριθμούνται, κατονομάζονται. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τέτοιου είδους πρόσωπα, απευθύνεστε σε εμά για να δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε. Μετά υπάρχουν οι περίφημες εταιρείες ε, θηρίδες εικονικές που είναι ενταγμένες σε ένα ε, ολόκληρο σύστημα για να μην ε, έχουν τους περιορισμούς ε, της χώρας έδρας και επιζητούν φορολογικούς παραδείσους. Πρέπει να σας πω ότι έκανα τη διατριβή μου για αυτό το θέμα ακριβώς πριν από 40 χρόνια και ξέρω μερικά πράγματα. Βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ ευρύ το θέμα. Δεν έχουμε έρθει αντιμέτωποι με αυτό γιατί στο δίκαιο ε, εμείς ασχολούμαστε με κάποιες υποθέσεις ε, που ε, έχουν εμφανιστεί από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ο νομοθέτης και μετά. Ο νομοθέτης όμως τώρα τι θέλει να κάνει. Είναι πολλές αυτές οι εταιρείε, οι ενδιάμεση και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θέλετε αυτές όλες να διωχθούν ή θέλει ο νομοθέτης να ε, ε, διώκει ε, τις εταιρείε αυτές που έχουν δημιουργηθεί συσταθεί μόνο για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και διαχείριση των κονδυλίων. Μετά υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν πέσει σε ένα σοβαρό επαγγελματικό σφάλμα. Έχουμε δεντολογικούς κανόνες, ρυθμίσεις, διοικητικές, κανονιστικές, εθνικές κλπ. Και κάτι άλλο που είναι και πιο ενδιαφέρον για μας είναι εκείνοι που έχουν ε, ε, λάθος εσφαλμένη συμπεριφορά. Ε, αυτό έχει να κάνει με την ε, επαγγελματική αξιοπιστία ε, του ενδιαφερομένου ή βαριά αμέλεια, παράδειγμα. Όταν προσπαθεί κάποιος να ασκήσει πίεση σε κριτικές επιτροπές, επιτροπές επιλογής ή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφαθμισμένων, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια που στα νομικά λέμε μέσον, έτσι ώστε να δούμε ποιοι συμμετέχουν σε περιπτώσεις δωροδοκίας ε, ε, ενεργητικής ή παθητικής. Ποιος πήρε μίζα, ποιος έδωσε. Γιατί δεν είναι ε, κάτι που έχει γίνει λάθος στην εκτέλεση της σύμβασης, αλλά είναι κάποια παράδεκτα πράγματα. Ορισμένοι προσπαθούν συστηματικά να αποφύγουν ε, όλα αυτά ε, αλλάζοντας διευθύνσεις και έχουμε κάποιες τέτοιες ε, περιπτώσεις ή, ή πλαστογραφούν τους λογαριασμούς τους στο ίντερνετ. Εμείς δεν μπορούμε να δράσουμε, όχι εμείς, όλος ο μηχανισμός και δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε. Και αν δεν κοινοποιήσουμε κάτι δεν έχει γίνει γνωστό και μπορεί να χρειαστεί χρόνια ολόκληρα. Και προσπαθούμε να εντοπίσουμε έτσι το βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα ή σφάλμα οι διατάκτες της Επιτροπής έχουν ε, πάρα πολύ αυστηρές εντολές, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται σε όλα τα άλλα θεσμικά όργανα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι κάθε τροποποίηση ή κάθε ε, απόπειρα ε, να ε, θολώσει τα νερά, ας πούμε, να κρύψει την ταυτότητά σου σε σχέση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι βαρύ επαγγελματικό σφάλμα. Όταν ο διατάκτης έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο ανάκτησης, ε, και θα επανέλθω σε αυτό γιατί η δουλειά μας δεν είναι ανάκτηση των κονδυλίων, τότε προσφεύγει σε εμά. Καλά, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ για το πώς ε, επιβάλλονται οι τιμωρίες και οι κυρώσεις κτλ. Ε, από εκεί έχουμε τις πληροφορίες μας. Από πού τις έχουμε? Από τους εσωτερικούς ελέγχους, από τις εσωτερικές έρευνες, από τις δράσεις της Όλαφ, από τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που δεν έχουμε λάβει πάρα πολλέ ακόμα, αλλά δεν αποκλεί τίποτα ότι μπορούμε να περιμένουμε και τέτοιες. Αυτό είναι ε, λοιπόν το κλασικό πλαίσιο για την παραβίαση των ε, σημαντικών υποχρεώσεων και τα σφάλματα. Λοιπόν, εδώ ε, ασχολήθηκα μέχρι τώρα με αυτά που εμείς ονομάζουμε πραγματική ε, ε, δικαιοδοσία του πάνελ, αλλά τι γίνεται με αυτούς που βρίσκονται ενώπιον του πάνελ και που βάσει συμβατικής σχέσης έχουν λάβει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι υπηρεσίες, είναι οι οργανισμοί, agencies και διάφοροι άλλοι οργανισμοί, αλλά βεβαίως και το ελεγκτικό συνέδριο, το δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, εάν ας πούμε η τράπεζα έχει πρόβλημα με έναν από τους ε, εργολάβους με τους οποίους έχει συμβατική σχέση για ένα από τα κτίρια της θα περάσει από αυτό το πάνελ. Ε, το καλό είναι ότι μέχρι τώρα ε, δεν ε, έχουμε άλλους συμβαλόμενους ε, από τις γενικές διευθύνσεις, ε, πολύ λίγο από τις υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. Μέχρι τώρα λοιπόν οι υπόλοιποι δεν έχουν απευθυνθεί σε εμά. Το πάνελ δεν είναι ένα στοιχείο άρρητα συνδεδεμένο με την Κομισιόν δεν ανήκει στην Κομισιόν δηλαδή. Είναι ανεξάρτητο το πάνελ και σας εξηγώ γιατί. Ε, πρόεδρος είναι ο υποφαινόμενος. Έχουμε πενταετή εντολή, μη ανανεώσιμη και ε, ε, στην ουσία ε, μη διαλυόμενη πριν από την εκνοή της προθεσμίας αυτής. Επομένως, εκ της φύσεώς μας είμαστε ανεξάρτητοι. Μας έχει ζητηθεί εξ αρχής να είμαστε ανεξάρτητοι. Υπάρχουν όμως ε, και ε, οι υπόλοιποι οι οποίοι εκπροσωπούν και υπάρχουν μετά οι υπόλοιποι διατάκτες τους οποίους δεν έχουμε δει και πολύ συχνά βέβαια είναι η αλήθεια και από τους οποίους ορίζουν οι υπόλοιποι ε, οργανισμοί. Ε, και ε, ε, έχουμε μαζί μας και την κυρία Βικτωρία Κασάδο η οποία είναι αναπληρώτρια του πλήρους μέλους που δεν είναι εδώ και έχουμε βεβαίως και τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της Κομισιόν που έχουν δυνατότητα να εδρεύουν στα Συμβούλια μαζί μας. Το πάνελ δημιουργήθηκε για να είναι ανεξάρτητο. Εμείς δημιουργηθήκαμε μετά από την απόφαση Planet. Ε, ε, ξέρετε την υπόθεση Planet, ε, είναι εταίρος. Υπήρχαν ήδη δυνατότητες δίωξης και μέσα δίωξης, όμως διαπιστώθηκε ορθώς ότι σε αυτές τις διαδικασίες οι οποίες έχουν κατασταλτικό χαρακτήρα, δεν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, διοικητική διαδικασία μεν, στην οποία να συμμετέχουμε, αλλά είναι κατασταλτικού χαρακτήρα και που σχετίζεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εμείς δημιουργηθήκαμε και γι' αυτό από όταν ανέλαβα ε, την ε, θέση μου ε, προσπάθησα έτσι ώστε τα δικαιώματα της άλλης, του αντίθετου μέρους να καλύπτονται, να έχει την δυνατότητα να αμυνθεί. Και βεβαίως οτιδήποτε και αν συμβαίνει το αντίθετο μέρος έχει δικαίωμα για τον πλήρη σεβασμό μας και την πλήρη δυνατότητα διαλεύκανσης από δική του πλευράς και υπεράσπισης υπεράσπισης ε, της υποθέσεως του. Δεν έχουμε όμως ε, ε, καμία δυνατότητα διερεύνησης και καμία δυνατότητα αυτόνομης κίνησης διαδικασίας. Και ε, μερικές φορές ε, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ε, αν πρέπει να ασχοληθούμε ή όχι. Ασχολούμαστε για να δούμε αν πραγματικά μπορούμε να συζητήσουμε την υπόθεση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα της άμυνας που μπορεί να έχει ή των αμυντικών εργαλείων που μπορεί να έχει ε, ο ενδιαφερόμενος. Λοιπόν, συνεδριάζουμε μία πρώτη φορά, εξετάζομαι ε, το αίτημα, βλέπουμε τα πραγματικά περιστατικά ε, και βλέπουμε τι νομική διαδικασία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Γιατί ελλείψη αποφάσεων τα πράγματα είναι είναι ασαφή. Εμείς περιμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξει δίωξη ε, δεν υπάρχει δηλαδή αναστολή δίωξης, απλώς περιμένουμε τι, θα, ε, τι θα αποφασιστεί. Ε, θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί εμείς δεν ανακατευόμαστε με τον δικαστή ανακριτή ή οτιδήποτε. Ε, βλέπουμε το συμβόλαιο και μελετούμε κτλ. Και, και αντί για τις 10 εργάσιμες ημέρες που ο κατηγορούμενος ή οι κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν και κυρίες οι οποίες δεν είναι πολύ καθαρές ε, στις διαδικασίες τους, ε, ε, ε αυτές οι 10 μέρες οι εργάσιμες έχουν γίνει πλέον 3 εβδομάδες, έτσι ώστε να δοθούν όλα τα εργαλεία και τα μέσα άμυνας για τον κατηγορούμενο η γραπτή διαδικασία όπου ο καθένας ε, βάζει και τη δικιά του ας πούμε πινελιά ε, είναι ο καλύτερος και σωστότερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται διαζώση σε αυτή τη διαδικασία, να πρέπει να, έχουμε μια ανταλλαγή συζητήσεων. Και εμείς λοιπόν καταλήγουμε σε ένα σχέδιο σύστασης το οποίο προωθούμε. Τώρα τελευταία είδαμε πολλούς εμπορευόμενους ε, που ε, ε αισθάνονται ε, κατηγορούμενοι απολύτως. Σε τέλη Δεκεμβρίου ας πούμε είχαμε μία δέσμη 30 σελίδων συν 50 σελίδες παραρτήματος όσον αφορά μία δίστροπη περίπτωση αμερικανικού δικαίου που έπρεπε να συζητηθεί μέσα Ιανουαρίου. Δεν μας άφηνε πολύ χρόνο αυτό. Εμείς εμβαθύναμε. και ε, Έχουμε ήδη 6-7 ζητήματα ενώπιον του, της ε, δικαιοσύνης για ένα πάνελ που, ισχύει, που λειτουργεί εδώ και πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Είναι ε, σημαντικό αυτό. Ε, ασχολούμαστε με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βεβαίως τα μέσα που έχουμε, ε, τι να σας πω, υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση να στείλουμε μηνύματα με το κινητό, δεν απαντάει ο ενδιαφερόμενος, στέλνουμε με ταχυδρομικά, δεν απαντάει ο ενδιαφερόμενος ε, τώρα, στέλνουμε το δικαστικό επιμελητή. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, εμείς δεν έχουμε σαν στόχο ε, να ξαναπάρουμε τα χρήματα, να ανακτήσουμε τα χρήματα τα οποία έχασε ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Αυτό που κάνουμε είναι να αποφύγουμε άνθρωποι που είναι επιζήμιοι με την έννοια ότι έχουν κλέψει εντό εισαγωγικών χρήματα ή προτίθενται να κλέψουν ή έχουμε βάσιμες υποψίες ότι προτίθενται και πρόκειται να κλέψουν αυτοί να βγουν εκτός κυκλώματος. Δεν έχουμε κάνει σαφείς υπολογισμούς, ξέρουμε. Και τι κάνουμε λοιπόν για να αποφύγουμε αυτούς τους επιζημίους ανθρώπους, τους αποκλείουμε ή ε, συνήθως ε, τους αποκλείουμε από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια, μερικές φορές κατ' εξαίρεση πέντε χρόνια. Αυτή τη στιγμή επίσης έχουμε και πλήρη δυνατότητα ε, οικονομικών προστήμων. Επιβολής δηλαδή οικονομικών προστήμων. Αν θέλετε μπορώ να σας πω και λεπτομέρειες Ε, υπάρχουν βέβαια μερικές περιπτώσεις που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί μπορεί να καταδικάσουμε κάποιον και να ε, ακυρωθεί αυτή η απόφαση και επομένως ε, ο εν λόγω κύριος να μην έχει πλέον κανέναν περιορισμό. Ε, κοιτάξτε, ε, ξέρετε ότι μερικές φορές εάν Εάν βάλει κάποιον, ε, του επιβάλλεις ένα οικονομικό πρόστιμο 30, 40, 100 χιλιάδες, μπορεί και να το πληρώσει. Αλλά εάν του επιβάλλεις αποκλεισμό τρίχρονο, μπορεί να σημαίνει ότι απλώς ε, θα πτωχεύσει. Και ακόμα χειρότερο είναι η ε, δημοσίευση. Η δημοσίευση είναι κατά κάποιο τρόπο η νέα εκδοχή της διαπόμπευσης. Αυτό που γίνεται λοιπόν με τη διαδικασία αυτή είναι ότι έχουμε κάποιου ανθρώπου που είναι επιζήτητε ζύμη δεν είναι οι καλύτερες δυνατές αναστροφέ, α το πούμε έτσι. Η δημοσίευση βεβαίως και δημοσιοποίηση είναι ε, πολύ δύσκολο θέμα. Ε, ε, εμείς αναφερόμαστε στην δημοσίευση, ε, καταδικάζουμε σε δημοσίευση η οποία υλοποιείται τρεις μήνες μετά την απόφαση γιατί πρέπει να δώσουμε στον αντίδικο όλες Όλες τις δυνατότητες, να ασκήσει δηλαδή κάθε δυνατότητα που έχει ενώπιον, να προσφύγει ενώπιον των δικαστηρίων. Ξέρετε ότι πάντα πρέπει να ε, προσπαθούμε να ισορροπούμε τις καταστάσεις όσο γίνεται περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε απλώς ε, να σφάξουμε στο γόνατο οποιονδήποτε έρχεται ε, μπροστά μας. Εμείς ε, είχαμε καταδικάσει ε, έναν ε, υποφορβέα ο οποίος ο δυστυχής ο οποίος είχε κλέψει 16.000 ευρώ. Το, το, το θέμα του ποσού δεν είναι πάντα πολύ σημαντικό, αλλά ξέρουμε Ξέρουμε ότι ε, σε ένα πολύ στενό περιβάλλον ε, του, του βγαίνει το όνομα ας πούμε η, ρετσινιά γιατί ξέρουμε ότι αυτός ε, ή ο άλλος έχουν εκλέψει. Ε, αλλά κάτι καινούριο τώρα που διαπιστώσαμε και είναι θετικό είναι τα διορθωτικά μέτρα. Μερικές φορές αυθορμήτως σταματάει. Σταματάει λέει το κράτος ότι εγώ τον έχω διώξει, τον έχω βγάλει από το κύκλωμα ε, αυτόν τον συγκεκριμένο. Τι να σας πω τώρα, ε, ε, υπάρχει και μία θεραπευτική πράξη η οποία, την οποία αναλαμβάνει ο διατάκτης σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά, αλλά πρέπει να πω η ε, επικύρωση, ε, συγγνώμη, η ακρόαση ή η, συμβου, παροχή ε, συμβουλής από τη δική μας πλευρά μπορεί να επισύρει την ακυρότητα της απόφασης και το λέω και λαμβάνοντας υπόψη και την το προηγούμενο λειτουργήμα που είχα εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. είναι, είστε πολύ γοητευτικός, είναι πολύ γοητευτικός ο λόγος σας. Ε, και σας ευχαριστούμε για αυτό. Ε, εδώ μιλάμε για το παλιό πάνελ, ε, το οποίο τώρα έχει συγχωνευτεί με το έντις, αλλά στο πάνελ πόσες υποθέσεις αντιμετωπίσατε για κακή συμπεριφορά, ας πούμε. Και στην βάση δεδομένων έντις πόσες είναι οι σημαντικές υποθέσεις. Αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση. Θέλει κάποιος να απαντήσει. Παρατηρήσει του κύριου Πενέρα εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι Parce que euh, la gestion de la Η διαχείριση της βάσης δεδομένων δεν είναι δική μου υπόθεση, είναι της κυρίας εδώ. Ε, από την άλλη όμως, να σας απαντήσω, 31 περίπου συνολικά συστάσεις απευθύναμε. Από τα τέλη του 2016 χρειάστηκε πολύ για να πάρει μπρο το σύστημα. Μετά υπήρξε μια μεγάλη διακοπή στα πλαίσια της έγκρισης και εν ώψη της έγκρισης του νέου δημοσιονομικού κανονισμού που άργησε, όπως ξέρετε, 31 είναι οι συστάσεις. Αν τα βρω στα χαρτιά μου εδώ, θα σας πω και περί τίνος πρόκειται. Τις περισσότερες ε, περιπτώσεις είναι παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων. nous avons des, des... Υπάρχουν έξι περιπτώσεις όπου πρόκειται για βαριά επαγγελματικά ασφάλματα. συνήθως αυτά θρίζονται. Γιατί είναι κλασικό στοιχείο το βαρύ παράπτωμα στην ε, δικαιοσύνη. Δηλαδή και να παραβιάσεις τη σύμβασή σου και αυτό βαρύ παράπτωμα είναι. 31 ε, που χρειάζονται το χρόνο τους και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που τις απορρίψαμε ως μη παραδεκτές ή κατά την εξέταση ο διατάκτης είπε «Ε, στο κάτω-κάτω το αποσύρω δεν αξίζει τον κόπο είναι μια παλιό περίπτωση. 31 συστάσεις είναι που είναι σε... έχουν πάρει το δρόμο τους, έχουν δρομολογηθεί για να δοθεί συνέχεια. Ωραία, θα συνεχίσω στα γαλλικά. Όσον αφορά την ε, πρώιμη ανείχνευση. Ε, είμαστε περιορισμένοι ε, όσον αφορά το χρόνο. Μπορούμε από τη στιγμή που ο διατάκτης μας ζητάει να κινηθούμε, έχουμε ένα χρόνο στη διάθεσή μας. Από το 2006 υπάρχουν νέες υποθέσεις. Μερικές σε ένα χρόνο, αν δεν έχουν περάσει από το πάνελ, έχουν αποκλειστεί, αλλά πολλές φορές εντωμεταξύ έχουν προσθεθεί επιπλέον πληροφορίες, αλλά ε, ε, σε όλα αυτά τα χρόνια. Ε, θέματα τα οποία μπήκαν, βγήκαν. Είχαμε περίπου 40 με 50, 50 θα έλεγα εγώ περισσότερο υποθέσεις και ελπίζω να απήντησα στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Αλλά υπάρχει κάπου ένα γραπτό κείμενο που αναφέρει αυτά που μας είπατε εδώ προσωπικά, κύριος Πενέρα. Ναι, αυτό τι να σας πω είναι θέμα της Κομισιόν, ωστόσο υπάρχει η έκθεση της Κομισιόν προς το Κοινοβούλιο για θέματα απάτη. Commission Staff Working Document, ε, το οποίο συνοδεύει το κύριο έγγραφο. Το πρώτο έχει ημερομηνία 20 Ιουλίου 2017 και έχουμε κι άλλο ένα της 3ης Σεπτεμβρίου 2018. Είναι απολύτως επίκαιρο λοιπόν. Δεν έχουμε για το 2016 γιατί ήταν αυτή η μεταβατική περίοδος. Έχουμε όμως τώρα ενδείξεις αρκετά συγκεκριμένες και όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούμε, ε, δηλαδή ανώνυμη καταγραφή και διαχείριση κτλ. Και όπως, ε, και όπως ε, είχαν μόλις και έλεγχο το, του εσωτερικού ελεγκτή, πραγματικά διαπιστώσαμε ότι ο Γενικός Υπεύθυνος είχε μεγάλη δυσκολία αντιμετώπιζε για να βρει την διεύθυνση του πάνελ. Η Γενική Διεύθυνση Μπίτζ ε, από ό,τι φαίνεται κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά μάλλον υπάρχουν άλλοι που δεν ενδιαφέρονται. Ξέρετε, αυτό προσθέτει δουλειά ε, και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μερικοί διατάκτες δεν θέλουν και να χώσουμε τη μύτη μας και να δούμε γιατί ε, άργησαν να αντιδράσουν. Και αυτό είναι μια στάση που, τι να σας πω, για να το πω πολύ χαλαρά, με εξέπληξε λίγο όταν τη διαπίστωσα, ε, γιατί εμείς τους βοηθάμε στην ουσία η απόφαση που παίρνει ο διατάκτης ε, συνήθως είναι το ακριβές αντίγραφο της σύστασης. Ε, όταν ε, ένας, δημοσιογρα... ένας, ένας υπάλληλος έχει μια μεγάλη ομπρέλα, την ώρα που αρχίζει να βρέχει θα την κλείσει. Πολύ ωραίο το παράδειγμά σας λέει η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πραγματικά ε, εδώ έχετε το κύριο έγγραφο του ΠΙΦ. Αυτό είναι ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ε, ωραία, τώρα ολοκληρώθηκε η δημόσια διαδικασία. Τελείωσε λοιπόν η δημόσια συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αν έχετε την καλοσύνη να αποχωρήσετε γιατί έχουμε μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Για τους υπόλοιπους θα συνεχίσουμε.